Alex. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, σαν απευθύνει το λόγο η πρόεδρος κυρία Κοράτσα Μπίλτ, ας ε, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε. Με μεγάλη μου χαρά σας καλασορίζω στη σημαντική και επίκαιρη αυτή συνάντηση, διότι τα παιδιά είναι τα πλέον ευάλωτα και αυτά που υφίστανται τα βαρύτερα προβλήματα από την κρίση του μεταναστευτικού μέχρι και 30 και 40% καμιά φορά ε, από αυτούς που έρχονται στην Ευρώπη είναι παιδιά και η Ευρώπη θα πρέπει να σημαίνει ασφάλεια για τα παιδιά. Είναι μάλιστα και επίκαιρη συνάντηση διότι μόλις είχαμε το φόρουμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύριο στην Μίνη Ολομέλεια έχουμε προφορική ερώτηση για τα αγνοούμενα παιδιά. Και ε, μάλιστα εμείς την ξεκινήσαμε αυτή την ερώτηση μετά από το συναγερμό που ε, χτύπησε πέρσι η ε, Ευρωπόλ. Έχουμε ε, συζητήσει πολύ εδώ για την τραγωδία των παιδιών που χάνονται εδώ στην Ευρώπη και την αποτυχία μας να τα βάλουμε σε ένα σύστημα προστασίας. Είμαστε εδώ διότι γνωρίζετε ότι στο Κοινοβούλιο επανεξετάζουμε ή αναθεωρούμε το πακέτο των μέτρων για το άσυλο και βεβαίως και άλλα συστήματα όπως το Eurodac και την οδηγία για την υποδοχή. Χρειάζεται πραγματικά να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας μαζί σας. Είναι κοινή ευθύνη μας και αναμένουμε βεβαίως τις ιδέες σας και ε, τις εισρωές από εσάς. Έχουμε ένα θαυμάσιο πάνερ, έχω τον Έντσο Μπιάνκο δίπλα μου, δήμαρχο της Κατάνια, στην Σικελία, Σικελία που βρίσκεται πραγματικά στα πρόσωπα του αγώνα. Καλώ ήλθατε. Ε, φροντίζετε για ασυνόδευτους ανηλίκους και παιδιά. Σας συγχαίρω για τις προσπάθειές σας και βεβαίως για τα όσα πράττει η Ιταλία για να σώσει ζωές στη Μεσόγειο. Έχουμε επίσης την Ματίνα Ερπ Κλούνεμαν, η οποία θα μας μιλήσει περισσότερο για την γερμανική προσέγγιση στο αγνώμενο ανήλικο η Γερμανία είναι από τις χώρες μέλη που έχουν υποδεχθεί τους μεγαλύτερους αριθμούς ανηλίκων και ασυνόδευτων παιδιών. Έχουμε τον κύριο Βερστάγεν επίσης, ίσως να μην λέω πολύ σωστά το όνομά σας, να με συμπαθάτε αν δεν το λέω καλά, που ε, χειρίζεστε το Ίδρυμα Πέραν λοιπόν των εθνικών πλαισίων, πάλι για το πολύ σημαντικό θέμα της κυδαιμονίας. Τέλος, τον κύριο Μαχμούντι από το Ένσα Κομάντε Φερμπούντ της Σουηδίας. Εσείς ο ίδιος υπήρξατε ασυνόδευτο, ασυνόδευτος ανήλικος. Σας επισκεφθήκαμε με επίσημη αντιπροσωπεία της ε, κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από το τεράστιο έργο που κάνετε από την βάση για να ε, δεχθείτε τα παιδιά και να φροντίσετε ώστε να μην είναι βάρος για την κοινωνία, αλλά να μπορεί να είναι πλούτος για την κοινωνία που τα υποδέχεται. Χωρίς λοιπόν άλλες καθυστερήσεις, πολύ ευχαρίστω να απευθύνω το καλό ορίσατε και στην Συμπρόεδρο, Κατρίνα Κινίτσι, την ε, Νάταλι Τζιμπεκ, τον, ε, ε, την, μάλλον, την Τζιν Λάμπερτ, συγκεντρώνουμε τις προσπάθειες ε, για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών. Το παιδί είναι πρωτίστως παιδί, ανεξαρτήτως από το, από το καθεστώς του ως μετανάστη ή οτιδήποτε άλλο. Και κάνουμε μεγάλη δουλειά εδώ στο Κοινοβούλιο για τη μετανάστευση. Τώρα λίγα πρακτικά, λίγες πρακτικές πληροφορίες. Όταν θα ακούσουμε όλους αυτούς τους εξαιρετικά ενδιαφέροντες ομιλητές, θα δώσουμε το λόγο στα μέλη στην αίθουσα. Παρακαλώ οι εθνικοί βουλευτές να ζητήσουν τον λόγο. Πρέπει να εγγραφείτε σε ένα χαρτί που θα λάβετε, ένα έντυπο που θα λάβετε από την γραμματεία. Για τους δικούς μας συναδέλφους ευρωβουλευτές αρκεί να σηκώσουν το χέρι τους. Θα σας δώσω τον λόγο για μέχρι δύο λεπτά. Αρχίζει τώρα η καταγραφή και θα σας πάρουμε τη σειρά που θα γραφτείτε. Χωρίς άλλες καθυστερήσεις, ο Έντσο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εξ ονόματος της ε, Επιτροπής ε, Περιφερειών. Είμαι δήμαρχος της ε, Κατάνια, είμαι πρόεδρος των Δήμων Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήμουν τυχερός γιατί ήμουν εισηγητής στην Επιτροπή Περιφερειών για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το δικαίωμα ασύλου και τη διεθνή προστασία. Ε, η πρόταση αυτή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε σαν στόχο να εναρμονίσει την κατάσταση και να εξομαλύνει τις ε, ανισότητες που υπάρχουν στο, στα εθνικά δίκαια όσον αφορά την, το δικαίωμα του, του ασύλου. Είμαι δήμαρχος ενός, ενός μεγάλου δήμου της Ικελίας που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της υποδοχής των μεταναστών που σώθηκαν από την ε, ε, ακτοφυλακή ε, της Ιταλίας, από το Ιταλικό Ναυτικό ε, στις ακτές μας ε, που προσπαθούσαν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές όταν κινδυνεύουν. Και όταν έχουμε γυναίκες και παιδιά που κινδυνεύουν να πεθάνουν και πολλοί ήδη έχουν πεθάνει ήδη, προσπαθούμε και θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να τους σώσουμε και είναι ε, κομμάτι βέβαια της διεθνούς, ε, του διεθνούς δικαίου αλλά και κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Βέβαια πρέπει να δούμε και ποια είναι η υποδοχή την οποία επιφυλάξαμε στα άτομα αυτά τα οποία ε, φτάσανε στις ακτές μας. Κάποιες ε, στιγμές ήμασταν τελείως μόλι. Το 2013, όταν ήμουν δήμαρχος ε, της Κατάνια, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση επίγουσα, αν θέλετε, επίγου, δραματική, διότι ούτε η χώρα μου ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί και έπρεπε ας πούμε να χρησιμοποιήσω όλους ε, τους ε, αθλητικούς χώρους ε, της πόλης μου και της περιοχής για να μπορέσω να φιλοξενήσω άτομα από το Αφγανιστάν, από την Σομαλία και από διάφορες άλλες χώρες που εξάγουν, αν θέλετε, μετανάστες και πρόσφυγες δεν θα πρέπει οι πόλεις ε, της πρώτης ε, εισόδου, αν θέλετε, να αναλαμβάνουν, να αναλαμβάνουν ε, τον, όλο το φόρτο της φιλοξενίας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.000 δήμοι και κοινότητα στην Ιταλία, σύμφωνα με ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζουμε, που φιλοξενούν τους μετανάστες ή τα άτομα στα οποία, στα οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα χορήγησης ασύλου. Τι πρέπει να κάνουμε, ε, προσπαθούμε να δούμε καταρχάς ε, ποια είναι η κατάσταση των ανηλίκων. Προσπαθούμε, προσπαθούμε αυτούς να προστατεύσουμε κυρίως, διότι έχει παρουσιαστεί μια φοβερή αύξηση των ε, μη συνοδευομένων ανηλίκων που έχουν φτάσει αυτές τις συγκελίες τα τελευταία χρόνια. Από τα 800 άτομα τα οποία έφτασαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία, ε, το 1 τέταρτο περίπου ήταν ε, ασυνόδευτοι, ασυνόδευτα ανήλικα. Το 1 τρίτο, συγγνώμη, περίπου. Ε, μάλλον, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο που να του συνοδεύει και να χάθηκε ή να μην έχει εμφανιστεί κτλ. Αλλά τέλο πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα ασυνόδευτα ανήλικα αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Θα πρέπει επομένως να ενδυναμώσουμε μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που δεν είναι ένα πρόβλημα ενός κράτους μέλους και δεν είναι κάτι παροδικό το οποίο σε ένα-δύο χρόνια θα εξαφανιστεί. Θα το αντιμετωπίσουμε και σε δύο και σε πέντε χρόνια το ίδιο πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία να ξεπερνάει το, το χαρακτήρα του κατεπήγοντος. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και με βάση την εμπειρία που έχουμε είναι η οικονομική παρέμβαση στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι οικονομικοί μετανάστες. Προφανώς αν είχαμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε σε αυτές τις χώρες, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες, χώρες προέλευσης, θα ήταν κάτι το θετικό. Επίσης κάτι άλλο, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την... Ε, ε, θα πρέπει να δούμε ε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις οργανώσεις που εποφελούνται οικονομικά από την παράνομη διακίνηση των ανθρώπων. Η εισαγγελία της πόλης μου, ε, της Κατάνιας, κάνει έρευνες για να μπορέσουμε να ε, φτάσουμε στα, να φτάσουν στα δικαστήρια ε, περιπτώσεις ατόμων που διακινούν διακινούν παράνομα ε, μετανάστες. Υπάρχουν, ε, έχουμε καταδικάσει άτομα τα οποία ε, ήταν υπεύθυνα για τον θάνατο πολλών ε, μεταναστών ε, που το μόνο τους έγκλημα ήταν ε, ότι αρνήθηκαν κάποια στιγμή να μεταφερθούν από, μια, από ένα μεγαλύτερο πλοίο σε ένα μικρότερο πλοίο. Και προφανώς το πλοίο βυθίστηκε. Επίσης, όπως σας είπα, επειδή έχει αυξηθεί ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων, πρέπει να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων. Στην ε, Επιτροπή Περιφερειών έχω ζητήσει να ε, ενισχυθεί ε, ο θεσμός του εγγυητή των δικαιωμάτων του ανήλικου. Και το τελευταίο θέμα είναι αυτό το οποίο αφορά στις πολιτικές ένταξεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, περί στην ε, πόλη μου είχαμε μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή, μεγάλη γιορτή του ε, καθολικού κόσμου. Η προστάτηδα της πόλης μου είναι η, η Σάντα Αγκάτα και είναι όντως μια πάρα πολύ ωραία γιορτή και ε, οργανώσαμε τις, ε, τους εορτασμούς ε, με μια ομάδα ανέργων της Κατάνια αλλά και μιας ομάδας ασυνόδευτων παιδιών έτσι ώστε ένας χώρος αποθήκευσης που είχε μείνει εγκαταλειμμένος να γίνει ένας, ένας μεγάλος κήπος. Και δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα, να, να αντιστρέψουμε μάλλον τον φαύλο κύκλο και να δημιουργηθεί κάτι θετικό. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει. Και σας ευχαριστούμε που μας επενθυμίσατε ότι είναι τα παιδιά μετανάστες που βρίσκονται σε κρίση και όχι εμείς και δεν είναι απλώς κρίση, είναι τραγωδία και εργαζόμαστε φυσικά και για την εφαρμογή της οδηγίας ε, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Και τώρα να περάσω αμέσως ε, στη δικαστή, στην κυρία Μαρτίνα Κλίνεμαν, Ερπ Κλίνεμαν, να μας ε, πείτε πώς χρησιμοποιείτε το αστικό δίκαιο για την προστασία των παιδιών. Η δικαστής κυρία Κλίνεμαν, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας για να σας αναπτύξω τα θέματα από την πλευρά του ε, ανθρώπου που ασχολείται στην πράξη με τα θέματα αυτά. Είμαι δικαστής σε δικαστήριο οικογενειακών θεμάτων. Γνωρίζετε ότι έχουμε υποδεχθεί πολλούς πρόσφυγες στην Γερμανία. Για την ώρα τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά στην Γερμανία είναι 55.000 περίπου. Τώρα, ποιος είναι ο ανήλικος. Ανήλικος είναι κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών ηλικίας. Το πρόσωπο αυτό έχει περιορισμένη ικανότητα συμβατική, δηλαδή να κάνει συμβάσεις. Ε, χρειάζεται την νομική εκπροσώπηση, την συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του για να μπορέσει ε, να ε, συμβληθεί. Αυτά τα γράφει ο αστικός μας κώδικας τα ανήλικα παιδιά συνήθως ε, βρίσκονται υπογονική γονική μέρημνα. Τώρα ποιο είναι ο ανήλικό. Ο ασυνόδευτο ανήλικο είναι ένα παιδί ανήλικο που δεν είναι εθνικός υπήκος και που εισέρχεται στη χώρα χωρίς παρουσία γονέως ή νόμιμου εκπροσώπου, νόμιμου κηδεμόνα. Το γερμανικό αστικό δίκαιο λέει ότι εφόσον κολλείονται οι γονείς από την άσκηση της γονικής μέρημνας, το Δικαστήριο Οικογενειακών Θεμάτων λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ανηλίκου. Το Δικαστήριο Οικογενειακών Θεμάτων έρει, αναστέλει την γονική μέρημνα στην περίπτωση όπου οι γονείς δεν έχουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα γονική μέρημνα και το δικαστήριο τότε διορίζει και μόνα. Αυτές είναι οι γενικές αρχές του γερμανικού αστικού δικαίου που εφαρμόζονται το ίδιο ακριβώ και σε εθνικέ υποθέσει όπω και σε διασυνοριακέ υποθέσει. Παντού εκεί ισχύει το αστικό δίκαιο. Μια άλλη άποψη για την οποία θέλω, μια άλλη πτυχή για την οποία θέλω να σα ενημερώσω είναι ότι τον Οκτώβριο του 2015 η διαδικαστική ικανότητα για να μπορούν να ζητήσουν άσυλο, η ηλικία δηλαδή η διαδικαστική ικανότητα, αυξήθηκε από τα 16 χρόνια στα 18. Γιατί έγινε αυτό σε μια στιγμή όπου φθάν, έφταναν στην Γερμανία τόσα πολλά παιδιά, γιατί αυξήθηκε η ηλικία διαδικαστικής ικανότητας. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι για να δοθεί έμφαση στην κυρίαρχη θέση των υπηρεσιών φροντίδας παιδιού και νεότητας. Αυτό σημαίνει ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος αντιμετωπίζεται πρώτα-πρώτα ως παιδί. Ένα παιδί το οποίο χρειάζεται προστασία. Ένα παιδί το οποίο χρειάζεται φροντίδα και βεβαίως χρειάζεται και εκπροσώπηση. Χρειάζεται έναν κηδεμόνα εφόσον μιλούμε για ασυνόδευτο ανήλικο. Ο εκπρόσωπος του παιδιού αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το παιδί και κατάθεση αιτήσεων ασύλου και άλλων, άσκηση των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στις διαδικασίες αυτές, δηλαδή συνοψίζοντας το ασυνόδευτο ανήλικο παιδί είναι πρώτα πρώτα ανήλικο παιδί και μετά αλλοδαπός. Εντυπωσιάστηκα σε διάσκεψη που ε, βρισκόμουν εδώ τον Δεκέμβρη γιατί νόμιζα ότι όλοι σκεπτόμαστε έτσι. Και τελικώς διεπίστωσα τότε ότι είμαστε, η δική μας κατάσταση στη Γερμανία δηλαδή είναι διαφορετική. Για μένα όμως ως δικαστήνα σε δικαστήριο οικογενειακών θεμάτων οι ορισμοί αυτοί είναι αυτονόητοι και για μένα είναι αυτονόητοι ότι τα ανήλικα παιδιά χρειάζονται και δαιμόνα. Έχουμε λοιπόν αυτομάτως μια παράλληλη προσέγγιση αφενός δηλαδή του αστικού δικαίου που φροντίζει να υπάρξει και η δαιμόνα του παιδιού, εκπροσώπησή του και από την άλλη μεριά ισχύει η νομοθεσία περί αλλοδαπών. Όταν οι κρατικές αρχές διαπιστώνουν ότι κάπου βρίσκεται ένα ανήλικο παιδί οπουδήποτε στη Γερμανία, τότε η τοπική αρχή νεότητας αναλαμβάνει την φροντίδα του παιδιού προσωρινά. Εντός μηνός γίνεται με την κατάσταση εντός της Γερμανίας και μετά η καινούρια τοπική αρχή νεότητας, αυτή δηλαδή που υποδέχεται το παιδί, αναλαμβάνει πλέον τη φροντίδα του. Ποιος εκπροσωπεί το παιδί στην αρχή, στην αρχική φάση, οι δύο τοπικές αρχές νεότητας εξουσιοδοτούνται από τον νόμο να δρουν ως εκπρόσωποι του παιδιού. πρώτον η τοπική αρχή νεότητας η οποία υποδέχεται το παιδί και μετά αυτή στην οποία ε, μεταφέρεται το παιδί, στην αρμοδιότητα της οποίας μεταφέρεται το παιδί. Και γενικά η δεύτερη αυτή η τοπική αρχή νεότητας ενημερώνει αμέσως το Δικαστήριο Οικογενειακών Θεμάτων. Τι κάνει το Δικαστήριο? Το Δικαστήριο ξεκινά την διαδικασία διορισμού και δαιμόνα όταν λάβει τη σχετική πληροφορία, κανονικά δηλαδή, από την αρχή νεότητας η οποία υποδέχεται το παιδί. Μπορεί να είναι διαφορετικό σε ορισμένες περιπτώσεις. Ορισμένες φορές μας ενημερώνουν οι συγγενείς του παιδιού. Άλλες φορές η τοπική αρχή νεότητας η οποία πρώτη υποδέχεται το παιδί και το λαμβάνει υπό την προστασία της. Μπορεί να μας ενημερώσουν για κάποια παιδιά τα οποία χρειάζονται κατεπηγόντως διορισμό και δε μόνος. Γενικώς πάντως έχει νόμι, νόημα να ενημερώνουν το Δικαστήριο Οικογενειακών Θεμάτων για το πότε έγινε η μετεγκατάσταση και είναι πλέον ξεκάθαρη η εγκατάσταση του παιδιού. Το Δικαστήριο Οικογενειακών Θεμάτων ακούει το παιδί, ακούει και τους γονείς, γιατί ορισμένε περιπτώσεις είναι δυνατόν να ακουστούν οι γονείς, διότι δεν είναι μακριά. Εννοώ δηλαδή ότι μέσω της τεχνολογίας είναι δυνατόν να ακουστούν. Ελέγχομαι βεβαίως και τα έγγραφα ταξιδιωτικά και άλλα που συχνά όμως δεν υπάρχουν και αυτό με οδηγεί να σας μιλήσω για ορισμένα προβλήματα που έχουμε, για παράδειγμα έλλειψη εγγράφων, ταυτοτήτων κλπ. που οδηγούν στο μεγάλο πρόβλημα της δυσκολίας εκτίμησης της ηλικίας. Είναι όντως ανήλικος ε, ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά μου. Το γεγονός ότι οι γονείς δεν μπορούν να ασκήσουν τη γονική μέρημνα για μακρό χρονικό διάστημα διότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι συχνά, πολύ συχνά, έχουν τακτική επαφή με τους γονείς τους, είτε βρίσκονται στη Συρία, είτε βρίσκονται στην Τουρκία, είτε αλλού. Έχουν όλοι κινητά τηλέφωνα και ε, κομπιούτερ. Αρκεί αυτό ώστε να θεωρηθεί ότι οι γονείς ασκούν τη γονική μέρημνα ή εκεί έχουμε την περίπτωση ότι κολλείονται να ασκήσουν τη γονική μέρημνα. Βεβαίως, εφόσον έχετε την επαφή μόνο με τεχνικά μέσα, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχουν την γονική μέρημνα. Μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους οι γονείς σε συγγενείς που ήδη κατοικούν στην Ευρώπη να ασκήσουν την κυδαιμονία του παιδιού. Αρκεί, τα, όμως αυτό στα μάτια του δικαστηρίου. Με μια απλή, ε, ε, απλή γραπτή εξουσιοδότηση Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, το Δικαστήριο Οικογενειακών Θεμάτων κηρύσσει την αναστολή της γονικής μέρημνας και διορίζει και δαιμόνα. Ποιος πληρώνει? Αυτός που υποβάλλει την αίτηση. Το δικαστήριο στην περίπτωση αυτή πληρώνει τους κηδεμόνες και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διορίζουμε συγγενείς αλλά διορίζουμε επαγγελματίες οι οποίοι αναλαμβάνουν το ρόλο του κηδεμόνος αυτοί οι κηδεμόνες από τη στιγμή εκείνη και μετά εκπροσωπούν το παιδί, τον Ασυνόδευτο ανήλικο, σε όλες τις διαδικασίες και περιπτώσεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις προοπτικές του. Να ζητηθεί άσυλο για το παιδί ή μήπως είναι καλύτερα να, ζητήσει, να γίνει αίτηση για έκτακτη άδεια για να μπορέσει να παρακολουθήσει εκπαίδευση ποιοι είναι οι λόγοι που είναι σημαντικοί για τις αρχές και που πρέπει να ενημερωθούν τα παιδιά. Δέχομαι την απόφαση που λαμβάνει η αρχή αλλοδαπών. Θα υποβάλω έφεση, αυτά είναι ερωτήματα για τον Κιδεμόνα. Αιτήσει για χρηματοδοτική υποστήριξη. Πολλών είδων αποφάσει. Μπορεί το παιδί να χρειάζεται ε, να υποστεί κάποια σημαντική εγχείρηση ή επίσης υπάρχουν έξοδα εκπαίδευσης. Όλα αυτά θα τα χειριστεί ο κηδεμόνας. Χρειαζόμαστε κηδεμόνες οι οποίοι να έχουν παιδαγωγικές ικανότητες αλλά και γνώση του πολιτιστικού ε, ιστορικού του παιδιού. Θα πρέπει να γνωρίζουν βεβαίως και το δίκαιο όλα και τους διαφορούς τρόπους εφαρμογής του για να μπορούν να εκπροσωπήσουν το παιδί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βεβαίω χρειάζονται και γλωσσικές δεξιότητες. Συνήθως δεν έχουν βέβαια τις γλωσσικές γνώσεις και χρειάζονται την παρέμβαση διερμηνέων. Εγώ βεβαίω μπορώ να σας πω μόνο τι γίνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Εγώ μιλούσα και με μία συνάδελφό μου στο Μόναχο που μου είπε ότι έχουν 400 διορισμούς κηδεμόνων την ημέρα. Δεν ξέρουν πια που να βρουν αρκετούς. Πάντως φαίνεται πως τα πράγματα βελτιώνονται στο μεταξύ και υπάρχουν περισσότερα πρόσωπα που είναι διαθέσιμα για να διοριστούν κηδεμόνες. Για την ώρα υπάρχει πάντως νομοσχέδιο, πρόταση η οποία συζητείται, ότι δηλαδή η τοπική αρχή νεότητας που υποδέχεται σε δεύτερη φάση το παιδί, υποβάλλει αμέσως αίτηση ασύλου. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι υποβάλλεται έγκαιρα η αίτηση. Αυτοί όμως που ασκούν κριτική στην ιδέα αυτή φοβούνται ότι η τοπική αρχή νεότητας που εκπροσωπεί το παιδί από την πρώτη στιγμή δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα για να τα πράξει αυτά. Δεν μου μένει πολύς χρόνος πια. Μία τελευταία λέξη λοιπόν για τους συνοδευόμενους ανήλικους και για αυτούς, για τα πρόσωπα δηλαδή, τα, που τα εκπροσωπούν εφόσον πρόκειται για γάμους ανηλίκων. Υπάρχει μια πρόταση νόμου να θεωρηθούν ανυπόστατοι οι, νο, οι γάμοι για πρόσωπα κάτω των 16 ετών και να θεωρηθούν τα παιδιά τα οποία είναι νυμφευμένα ή παντρεμένα τέλος πάντων κάτω 16 ετών ότι είναι ασυνόδευτα ανήλικα. Αυτό θα οδηγήσει σε μια βελτίωση, διότι θα μπορούμε να προχωρήσουμε ταχύτερα, να διορίσουμε κηδεμόνες με τις αναγκαίες ικανότητες και βρίσκω ότι είναι απολύτως σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά και κυρίως να τα προστατεύσουμε. Βεβαίως δεν είναι ποτέ απόλυτη προστασία, δεν είναι 100%, όμως είναι πραγματικά σημαντική και πλησιάζει το 100%. Σε ευχαριστώ πολύ ε, κυρία ε, Κλίνεμαν που μα εξηγήσατε ποιε είναι οι προκλήσει από τις πλευρά του δικαίου στη Σουηδία. Έχουμε πάνω από 100 κορίτσια που μας ήρθαν ε, παντρεμένα και μάλιστα ορισμένα έχουν και παιδιά. Πρόκειται για πραγματικά μια τεράστια πρόκληση για το δίκαιο και οι διάφορες τοπικές κοινότητες αναζητούν τρόπους να το αντιμετωπίσουν και χρειάζεται ασφαλώς ασφάλεια δικαίου για το πώς θα αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις αυτές. Τώρα για την κυδαιμονία θα δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Βερστέγγεν που είναι ο Γενικός ε, Μάνατζερ του Ιδρύματος Νίγενς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι με τιμά ιδιαίτερα που μπορώ να σας πω για το σύστημα επιτροπίας ε, στην Ολλανδία. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο το πιστεύουμε, δεν θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί. Το NIDOS ε, είναι ένας φορέας επιτροπίας ε, ε, σήμερα παρέχει επιτροπία 6.000 περίπου ασυνόδευτους ανηλίκους. Εμείς μπορούμε σήμερα να χειριστούμε 6.000 παιδιά πριν να χρόνο είχαμε 3.000 παιδιά παραπάνω από ό,τι στο παρελθόν και πάλι τα καταφέρναμε. Θα σας εξηγήσω πώς. Το 85% των παιδιών μας προέρχονται από χώρες που βρίσκονται σε πόλεμες σειράξεις από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και από την Ερυθρέα. Το 85% των παιδιών μας δηλαδή. Επομένως δεν είναι οικονομικοί μετανάστες και χρειάζονται όλη προστασία. Πώς λειτουργεί το σύστημα στην Ολλανδία. Θα σας πω και για την Ευρώπη, γιατί προσπαθούμε να συνεργαστούμε με άλλα ιδρύματα επιτροπίας στην Ευρώπη. Και μαζί καλύπτουμε τις οργανώσεις NGI. Μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. NGI.eu Λοιπόν, υπάρχει και το θέμα του ορισμού. Δηλαδή μπορώ να σας εξηγήσω τι σημαίνει επιτροπή στις κατοχώρες, αλλά τι σημαίνει επιτροπή σε άλλες χώρες. Αυτό διαφέρει. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό ορισμό λοιπόν για τον όρο επιτροπή, guardianship και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια σχέδια κειμένου. Ορισμό στην Ολλανδία. Θα σας δώσω αυτόν τον απλό ορισμό εργασίας, ότι είσαι υπεύθυνο αλλά και λογοδοτής για την ευημερία των παιδιών που έχεις αναλάβει. Και τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε εξουσίες, αρμοδιότητες ως γονείς, αλλά λογοδοτούμε και ως γονείς. Έτσι λοιπόν πράγματι πρέπει να τα φροντίσουμε αυτά τα παιδιά. Δεν μιλάμε μόνο για νομική εκπροσώπηση, αλλά και για φροντίδα. Πρέπει να φροντίσουμε την υγεία τους, την εκπαίδευσή τους, ε, τις νομικές διαδικασίες. Είμαστε υπεύθυνοι για όλα αυτά που γίνονται και πρέπει να γίνονται με έναν σωστό τρόπο και αυτά όλα πρέπει να τα κάνουμε εμείς και τα διαχειριζόμαστε. Τώρα για τον Ίντους κάτι ακόμη. Είμαστε ανεξάρτητο φορέα, είμαστε μη κυβερνητική οργάνωση, πληρώμαστε από την κυβέρνηση και παρόλα αυτά μπορούμε να είμαστε μη κυβερνητική οργάνωση. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ανεξάρτητο φορέα επιτροπίας, γιατί ενίοτε το συμφέρον του παιδιού Ε, ουσιαστικά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ποιος είναι ο αρμόδιος, η κυβέρνηση ή όχι. Μας διορίζει ένας δικαστής ε, που βοηθά. Ένα παιδί λοιπόν που είναι στις κάτω χώρες χωρίς τους γονείς του χρειάζεται έναν επίτροπο. Μας διορίζει λοιπόν ε, δικαστής ε, και στο αστικό δίκαιο ορίζεται τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να φροντίσουμε την κατάλληλη ανάπτυξη του παιδιού. Και αν κινδυνεύει η κατάλληλη ανάπτυξη του παιδιού, θα πρέπει να παρεύουμε. Και αυτό κάνουμε και μας βοηθά ότι είναι καταγραμμένο αυτό στην νομοθεσία γιατί η πολιτική και ο νόμος δεν είναι πάντοτε το ίδιο. Έτσι λοιπόν αυτό μας βοηθά να είμαστε σε ισχυρή θέση για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του παιδιού. Επίσης μας εποπτεύουν κιόλας. Πρόκειται λοιπόν για ένα φορέα επιτροπίας. Σήμερα 600 άτομα εργάζονται στον Ίντος και μας ε, εποπτεύει η επιθεώρηση νεολαίας. Και πρέπει να είμαστε επαγγελματικά οργανωμένοι, έχουμε ένα πιστοποιητικό, κάθε χρόνο πρέπει η Επίτροπή μας ε, ως δικηγόροι να καταρτίζονται, να μελετούν κτλ. Είναι όλοι επαγγελματίες, είναι ε, άνθρωποι που έχουν πτυχίο, είναι κοινωνική λειτουργή και προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των παιδιών αυτών και των παιδιών που έχουν την Ολλανδική υπηκότητα και προσπαθούμε να θετήσουμε και μεθοδολογία είναι το σημαντικό, ότι δεν λειτουργεί μόνο σου. Λαμβάνει πάρα πολύ σημαντικέ αποφάσει για ένα παιδί, αλλά αυτό γίνεται ομαδικά και εποπτεύεσαι από τον διευθυντή σου, υποστηρίζεσαι από τους συναδέλφους σου ή από ψυχολόγους από την οργάνωση. Δεν ζεις λοιπόν μέσα σε μία φούσκα. Και επίσης υπάρχουν ε, και ανταλλαγές διδαγμάτων ο ένας μαθαίνει από τον άλλο, ακούς από τον συνάδελφό σου, μαθαίνεις από τον συνάδελφό σου ότι ίσως αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, θα σε διορθώσει ο συνάδελφος για να το κάνεις καλύτερα. Τώρα για το σύστημα και τη θέση του επιτρόπου στο σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να σα το εξηγήσω εδώ. Στις κατοχώρες είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Θα σα εξηγήσω λοιπόν. Υπάρχει μια οργάνωση επιτροπή για συνόδευτου ανηλίκους για το σύνολο τη χώρα, Ένα παιδί που φτάνει στις κατοχώρες και θα ζητήσει άσυλο, θα πρέπει να πάει σε ένα κέντρο κατάθεση τη αίτηση. Είναι στο βορρά, πάρα πολύ δύσκολο να το βρει κανεί. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν και καταθέτουν την αίτηση ασύλου και την πρώτη στιγμή που φτάνουν εκεί, την πρώτη μέρα θα, συναντήσουν ήδη, θα συναντηθούν ήδη με τον επιτροπό τους. Και αυτό σας το εξηγώ, γιατί ίσως σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία μπορεί να μιλάβει αυτό χώρα την πρώτη μέρα, μπορεί να συναντήσει το παιδί, τον επίτροπο αργότερα. Εμείς τώρα τι μάθαμε. Ότι τα κορίτσια από την Ιγυρία που έρχονται στις κάτω και ζητούν άσυλο, όλα καταλήγουν ε, σε πορνεία, όχι μόνο στις κατοχώρες αλλά και στο Βέλγιο, στην Ιταλία και αλλού. Και το Υπουργείο, ε, μάλλον ο Υπουργός ε, που ήταν υπεύθυνο για αυτό το θέμα, ρωτήθηκε από το Κοινοβούλιο τι κάνετε γι' αυτό και είπε εγώ δεν είμαι υπεύθυνο, ήρθε λοιπόν σε εμά και είπαμε εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Αλλά στον τύπο ε, είχε και γραφτεί ότι αυτά τα κορίτσια εκπορνεύονταν στο Βέλγιο και είχαν εξαφανιστεί όλα αυτά τα κορίτσια πριν να διοριστεί επιτροπός για αυτά. Έτσι λοιπόν σήμερα από την πρώτη στιγμή διορίζουμε τον επίτροπο γιατί τα παιδιά είναι ε, ευπαθή και βλέπουμε ποια παιδιά είναι ευάλωτα, ποια παιδιά μπορεί να είναι θύματα εμπορία και από την πρώτη στιγμή παίρνουμε μέτρα. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που είναι κάτω από 15 ετών όλα θα τεθούν σε θετέ οικογένειε κατευθείαν από το κέντρο κατάθεση τη αίτηση ε, και θα είναι οικογένειε ε, από την ίδια, από την ίδια κουλτούρα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, έχουμε ειδικά κέντρα προστασίας ε, για τα παιδιά αν μπορεί να είναι θύματα εμπορίας. Μπορεί, παραδείγματο χάρη, ε, να έχεις ένα πρόβλημα και να σε βοηθήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, θα το εξηγήσω και ενδιαφέρει η δική μας μέθοδος από τις άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν ήδη υπάρχει ένας επίτροπος για να δει ποια παιδιά είναι ευάλωτα και πού θα πάνε από εκεί και πέρα. Είναι στα σύνορα αυτός ο Επίτροπος. Λοιπόν, μπορεί να πα, το χάρη, σε ένα κέντρο για του ασυνόδευτε ανηλίκου, σε ένα μεγάλο κέντρο. Αυτό δεν μα αρέσει, θέλουμε να το αλλάξουμε. Αυτό συμβαίνει του πρώτου μήνε που φτάνει το παιδί στι κατοχώρε και καταθέτει την αίτησή του για άσυλο ετοιμάζεσαι από το δικηγόρο ως παιδί, θα υπάρξουν και κάποιες ιατρικές εξετάσεις και στο τέλος του μήνα θα καταλάβεις αν μπορείς να μείνεις στις κατοχώρες ή όχι, αν μείνεις, αν μπορείς να μείνεις όμως ο Επίτροπος θα φροντίσει το επόμενο στάδιο της παραμονής σου στις κατοχώρες και τότε θα, είτε θα πας σε θετή οικογένεια είτε θα σου δώσουν ε, ε, κάποια στέγη. Ο Επίτροπος θα φροντίζει ότι θα βρει το σωστό μέρος για να κατοικήσεις ή θα παρέμβει αν θεωρεί ότι τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει και θα δει πώς αναπτύσσεσαι ως παιδί. Κάθε μήνα βλέπουμε αυτά τα παιδιά που μένουν, συζητάμε μαζί τους για το πώς τα πάνε, βλέπουμε τι γίνεται με το σχολείο τους, με την υγεία τους και αν χρειάζονται αλλαγές παρεμβαίνουμε. Αυτά όλα γίνονται από επαγγελματίες που ξέρουν ε, πώς ε, μπορούν να λειτουργήσουν και να εργαστούν με αυτά τα παιδιά γιατί έρχονται από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Θα ήθελα να σας πω κι άλλο, αλλά βλέπω ότι έχει τελειώσει ο χρόνος μου. Τι χρειάζεται τώρα. Λοιπόν, Κάθε παιδί θα πρέπει να έχει έναν ανεξάρτητο επίτροπο με εμπειρία. Νομίζουμε ότι είναι καλύτερο να είναι και επαγγελματία ο άνθρωπο αυτό. Και κάθε μεταγκατάσταση τοποθέτηση παιδιού θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού καταρχήν και το παιδί καταρχήν θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί σε μια οικογένεια και αν όχι σε κάποιο ειδικό κέντρο. Και όσο πιο μικρή είναι η δομή, τόσο το καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω ε, να μπορέσετε και εσείς όπως και η δικαστής Μαρτίνα να διαθέσετε το υλικό που έχετε στους συναδέλφους γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πριν δώσω το λόγο στον Ομαν θα ήθελα να ε, ρωτήσω αν κάποιος έχει να κάνει κάποια ερώτηση στον κύριο Μπιάνκο. Μόνο στον κύριο Μπιάνκο, διότι πρέπει να φύγει, δυστυχώς. Άρα, ρωτώ, συνάδελφοι, έχετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Μπιάνκο, η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, κύριε Ένσο Μπιάνκο. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση για αυτό το οποίο υπογραμμίσατε και συγχαρήκατε γενικότερα την, τις όλες τις προσπάθειες τις οποίες, οι οποίες γίνονται για την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών ε, πολιτικών και των νομοθεσιών. Όμως είναι δίκοπο μαχαίρι αυτή η εναρμόνιση. Γιατί αν δείτε πώς γίνεται η εναρμόνιση των νομοθετικών κειμένων, κανονισμών οδηγιών κτλ, η εναρμόνιση γίνεται προς τα κάτω. Δεν είναι, δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε δηλαδή βέλτιστες πρακτικές ή καλύτερες πρακτικές στα κράτη-μέλη. Αναφέρομαι ε, στα, στην οδηγία για τα προσόντα, όπου η, η, διάρκεια ε, για την χορήγηση ε, ασύλου μέσα στα πλαίσια της οδηγίας για την χορήγηση του ασύλου αναφέρεται η περίοδος ενός έτους ενώ σε υπάρχουν χώρες όπου εφαρμόζεται πολύ ε, λιγότερος ο χρόνος, ακόμα και στην Ιταλία. Όταν μιλάμε για τις ελάχιστες απαιτήσει ε, για τη χορήγηση του ασύλου, γίνεται πάντα η εναρμόνιση προς τα κάτω και μπορεί να ανασταλεί και η προστασία και ε, επανεξετάζεται με βάση των καταλόγων ε, των ασφαλών χωρών που δεν είναι ποτέ όλες ασφαλείς και αυτοί οι κατάλογοι είναι είτε ευρωπαϊκοί είτε εθνικοί. Ε, πολύ σωστά ε, επίσης ε, χαίρεστε διότι ακριβώς και το Ιταλικό Ναυτικό και η Ακτοφυλακή έχουν κάνει ε, τεράστιες προσπάθειες για την διάσωση των μεταναστών ε, στις Ιταλικές ακτές. Ο διευθυντής όμως της Frontex είπε ότι αυτές οι επιχειρήσεις διάσωσης ε, που εκτελούνται από μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα σταματήσουν και δεν θα συνεχιστούν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του λαθρεμπορίου. Τι έχει να πείτε γι' αυτό όντως μίλησα για την εναρμόνιση που πρέπει να αποτελεί ένα θετικό στόχο και υπογραμμίζω πώς. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι ε, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το άσυλο ή όχι, να είναι διαφορετικά στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κράτη τα οποία αναγνωρίζουν το δικαίωμα ασύλου στους ε, Σύριους ή στους Αφγανούς, ενώ άλλες χώρες όχι. Ε, άρα χρειάζεται περισσότερη εναρμόνιση εδώ και αυτό είναι θετικό. Τώρα, τα σημεία τα οποία αναφέρετε εσείς, ε, τις, απε, τις ελάχιστες απαιτήσει, ε, η διάρκεια και τα λοιπά, των διαδικασιών κτλ. Όντως ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και στην, στην Επιτροπή Περιφερειών και μετά και από δική μου πρόταση και είπαμε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις διαφορές αυτές. Δηλαδή η εναρμόνιση είναι θετική γενικά, πρέπει όμως η εναρμόνιση να είναι ένα εξελικτικό, μια εξελικτική διαδικασία και όχι μια ε, περιοριστική. Στην Κατάνια, στην πόλη μου, σε ένα δημοτικό κτίριο φιλοξενούμε την, ε, μια επιχειρησιακή έδρα της Frontex, αλλά και άλλες ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες υπεύθυνε για τα θέματα αυτά της μετανάστευσης, όπως η Europol. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εάν η Frontex ήταν, ήταν στην Πολωνία, με όλο το συμβασμό που τρέφω στην Βαρσοβία ή στην Πολωνία, θα έλεγα ότι ε, η Frontex πρέπει να είναι εδώ, όχι εκεί. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις διάσωσης να γίνονται στην, στα χωρικά ύδατα της Λιβύης και υπάρχουν κάποιες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που φτάνουν ε, στις ακτές της ε, Λιβύης ακόμα. Και αυτό βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο, που κάνει πιο εύκολη όχι την διάσωση αλλά άλλου είδους επιχειρήσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται η διάσωση στη θάλασσα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει βήματα προόδου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις οργανώνουν την αναχώρηση των μεταναστών με γραφεία ε, από την Λιβύη και με την ε, διάσωση στα χωρικά ύδατα της ε, Λιβύης. Αυτή δεν είναι διάσωση, αυτό είναι κάτι άλλο προσωπικά την, θα, θα έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε να έχουμε κάποιες οργανώσεις σε κάποιες χώρες να δημιουργηθεί ένας ανθρωπιστικός διάδρομος ε, δηλαδή. Δηλαδή αυτοί που έρχονται από χώρες ε, που όντως ε, δικαιούνται την χορήγηση του ασύλου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποιες διαδικασίες που να τους καθιστούν ασφαλείς. Δηλαδή να υπάρχει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπιάνκο. Ε, ζητά από όλους να τον χειροκροτήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Ε, τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπε. Να σας πω ότι ε, πέρυσι ε, ε, οργανώσαμε μία επίσκεψη στην Λαμπεντούζα. Ε, Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα προβλήματα υπάρχουν διότι δεν υπάρχουν ε, πολλές πρωτοβουλίες κατάσταση και μεταφοράς των ε, μεταναστών. Ε, δηλαδή πιστεύω ότι η νομοθεσία υπάρχει, δεν εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ομίντ Μαχμουντή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και που μου δίνετε και τη δυνατότητα να τοποθετηθώ και να αγωνιστώ για να ζούμε όλοι σε μια μεγάλη κοινότητα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Έρχομαι από το Αφγανιστάν και ανήκω σε μια εθνοτική ομάδα στους Αζάρους. Βρίσκεται στα σύνορά μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν. Ήταν ε, πολύ δύσκολο τότε να ζήσει κανείς εκεί. Κυκλοφορούσαν πάρα πολύ ένοπλοι και ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέχρι και να βρεις ένα πακέτο τσιγάρα. Ήταν ε, πολύ μεγάλη επιτυχία για μένα που κατόρθωσα να φύγω. Λέγομαι ο Μίτ Μακμούντι, είμαι από το Αφγανιστάν. Έφτασα στη Σουηδία το 2011 και κατόπιν έγραψα ένα βιβλίο που λέγεται «Η αθώοι εγκληματίες και περιέγραψα γιατί έφυγα από τη χώρα καταγωγής μου, πώς έφτασα στη Σουηδία και πώς εγκαταστάθηκα στη Σουηδία. Στη συνέχεια άρχισα να σκέφτομαι τα παιδιά που έρχονται μόνα τους, ασυνόδευτα και φυσικά μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πάρα πολλές εμπειρίες ζωής, πολύ διαφορετικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε παιδιά που έρχονται από πάρα πολλές χώρες, από 82 διαφορετικέ χώρε το χάρη και προσφέρουν λοιπόν 82 διαφορετικές εμπειρίες στη Σουηδία. Έτσι λοιπόν ε, ήθελα να δημιουργήσω μια οργάνωση και έτσι δημιούργησα τη Σουηδική Οργάνωση για του Ασυνόδευτους Ανήλικου, στην ε, SM Condes Forbund. Όμως ε, βλέπαμε ότι υπήρχαν λιγότερα κορίτσια από ότι αγόρια που έρχονταν στη Σουηδία. Ρωτήθηκα γιατί και έτσι λοιπόν ε, έγραψα και το δεύτερο βιβλίο μου που επικεντρώνεται σε αυτό το θέμα στη συνέχεια. Ε, εργάστηκα σε, επί ενός ντοκιμαντέρ και δημιούργησα και μια επιχείρηση για να έχουμε ένα μεγαλύτερο αντίκτυπο στη Σουηδική κοινωνία αυτή η επιχείρηση ουσιαστικά φορούσε τη διάδοση ιδεών, ένα κέντρο για τη διάδοση ιδεών, εργάστηκα πέντε χρόνια σε αυτό τον τομέα. Έτσι λοιπόν, ένας ε, πρόσφυγας ε, νέος που έφτασε πριν 5-6 χρόνια μπορεί να φτάσει στη θέση που είμαι σήμερα. Κάποιος που φτάνει στη Σουηδία ήδη την επόμενη μέρα αρχίζει να μπορεί να βοηθά τη Σουηδία η Ένωση μας ε, την Ένωση μας τη διαχειρίζονται οι ίδιοι νέοι. Ο στόχος μας είναι να ακουστούμε. Θα πρέπει οι νεοφυχθέντες να μπουν το συντομότερο, να ενταχθούν το συντομότερο στην κοινωνία για να μπορούν να συνεισφέρουν. Μακροπρόθεσμα θέλουμε να δημιουργήσουμε και τοπικές ε, οργανώσεις για να καλύψουμε το σύνολο της Ιουδικής Επικράτειας. Σήμερα έχουμε Μάλιστα, μάλλον ο στόχος ήταν να δημιουργήσουμε πέντε τοπικά κέντρα, σήμερα έχουμε φτάσει στα 16. Τι σημαίνει αυτό. Ότι θέματα όπως... Ε, ότι μάλλον ε, μπορούν οι νέοι να είναι αντικείμενο θερμής υποδοχής και να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία. Τι βλέπουμε ότι υπάρχουν εδώ δύο άνθρωποι, εγώ και άλλος ένας συνάδελφος που είναι εδώ στην αίθουσα. Φτάσαμε ως ασυνόδευτοι ανήλικοι στη Σουηδία. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι να γίνονται αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να ακουστούν, να γίνονται δεκτοί, να μπορούν να μιλήσουν για την κατάστασή τους. Το 2011 όταν έφτασα στη Σουηδία με έβαλαν μαζί με άλλους 700 νέους ε, σε ένα κέντρο. Σήμερα οι άνθρωποι αυτοί έχουν ε, γίνει δικηγόροι, οδοντίατροι. Βλέπετε τον κατάλογο εδώ. Δεν υπήρχαν ε, κορίτσια στο κέντρο εκείνο, μόνο αγόρια ήμασταν. Αποτελούμε λοιπόν καταρχήν ένα μεγάλο πόρο για μας τους εαυτούς μας καταρχήν, αποτελούμε και πόρο και για την κοινωνία. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται ότι είμαστε βάρος, ότι είμαστε άχθος. Όμως ε, στις ε, σκανδιναβικές χώρες ε, χρειάζονται μετανάστες για να υπάρχει μια βιώσιμη κοινωνία. Στη συνέχεια βλέπουμε διάφορες κατηγορίες ανθρώπων που καταφτάνουν. Όταν κάποιος είναι νέος, θέλει να ξεφύγει από τις τρομοκρατικές ε, ομάδες, από τον πόλεμο. Όσοι δεν μπορούν να φύγουν, δυστυχώς ε, μπορεί να βρουν και το θάνατο στις ε, χώρες καταγωγής τους. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται ο πόλεμος. Στο Αφγανιστάν μια τελευταία μελέτη μας δείχνει ότι το 50% των ε, κοινοτήτων δικούνται από τρομοκράτες. Στη συνέχεια Υπάρχει και ο στόχος του να σώσει τη ζωή ενός άλλου. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για να σωθούν. Οι τρομοκράτες ε, λένε ότι αν σκοτώσεις ε, κάποιον θα πας ε, στον παράδεισο και αν σκοτώσεις π.χ. χάρη 21 άτομα τότε θα πάνε και γονείς σου στον παράδεισο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κανείς δεν θα φεύγει από τη χώρα του <laughs> για ευχαρίστηση. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Στο Αφγανιστάν έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια πόλεμο που θαρίζει Μέχρι σήμερα ο πόλεμος θερίζει. Δολοφονήθηκε και ο βασιλιάς από τους Σοβιετικούς και περίπου 63% των Αζάρων έφυγαν στο Ιράν. Εκεί έπρεπε να ζήσουν σε φρικτές συνθήκες, δεν γίνονταν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και φύγαμε από το Ιράν και μπήκαμε στο Αφγανιστάν για να γλιτώσουμε από τον ρατσισμό. Εκεί υπήρχαν πάλι τεράστιες διακρίσεις μας συμπεριφέρονταν σαν προδότες της πατρίδας. Και πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς ήρθαν στην Ευρώπη το 2015-2016 για να ζήσουν με έναν εξωπρεπή τρόπο. Οι άνθρωποι αυτοί διανύουν το Ιράν για να έρθουν στην Ευρώπη. Όμως ε, στο Αφγανιστάν υπάρχουν ειδικοί κώδικες για να μπορεί κάποιος να επιβιώσει, θα πρέπει να ξέρει, να αποφεύγει τους τρομοκράτες, ε, τους παιδεραστές, διάφορες απειλές. Πραγματικά θα πρέπει εκεί να επιστρατεύσει όλες τις ικανότητες για να γλιτώσει. Και ή πρέπει να φύγεις γιατί δεν μπορείς να επιβιώσεις ή θα μπει σε τρομοκρατική ομάδα. Και οι άνθρωποι φεύγουν για να μπορούν να βρουν δουλειά και να μπορούν να στείλουν ε, κάποια χρήματα στην οικογένειά τους, για να επιβιώσει η οικογένειά τους. Έχουμε και τέτοιους ανθρώπους. Ε, τώρα εδώ σας αναφέρω διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Ε, όλοι ήταν όμως σε δύσκολες καταστάσεις. Όταν έφτασα για πρώτη φορά στη Σουηδία, είχα ένα στόχο. Ο στόχος μου ήταν να πάρω με άδεια παραμονής εργάστηκα, σπούδασα, ήθελα πράγματι να ενταχθώ στη Σουηδική κοινωνία. Και μετά, αφού πήρα την άδεια παραμονής, ήθελα να δημιουργήσω μια επιχείρηση, ήθελα να δημιουργήσω μια οργάνωση, ήθελα να βάλω τα δυνατά μου για να συνεισφέρω στη Σουηδική κοινωνία. οι νόμοι που μπλοκάρουν τους ετούντες άσυλο είναι προβληματικοί. Γιατί ουσιαστικά δεν επιτρέπουν την χορήγηση μόνιμης άδειας παραμονής. Αυτά από μένα και θα σταματήσω εδώ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συνεισφέρετε στην συζήτησή μας και γιατί ακριβώς μας μεταφέρετε όλη την ενέργειά σας στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Ε, Είσαστε ζωντανή απόδειξη ότι μια οργάνωση μπορεί να επιβιώσει και εσείς προσωπικά έχετε αυτή την θέληση να συνεισφέρετε στην ε, εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και στην διάσωση των παιδιών. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Λόρδο Σόλι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ εντυπωσιακά όλα ακούσαμε. Πολύ χρήσιμα. Μία ερώτηση όσον αφορά τους κηδεμόνες. Από πού επιλέγονται οι κηδεμόνες. Είναι επαγγελματίες ε, ή προσλαβαίνετε κάποιους ανθρώπους ε, από κάπου και τους εκπαιδεύετε. Και μετά ένα σχόλιο στον κύριο Μαμούντι ε, που πραγματικά τη μαρτυρία του τη βρήκα συγκλονιστική. Ε, στην ε, Βουλή των Λόρδων δημοσιάσαμε μία έκθεση για τα συνόδευτα παιδιά και είχαμε διάφορες μαρτυρίες. Μία από αυτές από ένα παιδί που προερχόταν από το Αφγανιστάν και είχε ζήσει διάφορες τραυματικές εμπειρίες. Ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι είναι δύσκολο για ανθρώπους που ζουν σε μία χώρα που λειτουργεί κανονικά να συνειδητοποιήσουν ε, το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που προέρχονται από χώρες σαν το Αφγανιστάν. Ε, και επειδή σε κάποιες ε, περιοχές είναι, θεωρείται ασφαλής χώρα το Αφγανιστάν, κάποια από αυτά τα παιδιά μπορούν, τα αγόρια μπορούν να επιστρέψουν στην χώρα τους. Τους επιστρέφουμε στη χώρα τους και υπάρχει ο κίνδυνος είτε να ε, τους ε, πάρουν οι Ταλιμπάνα ή να τους τιμωρήσει η οικογένειά τους. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ε, υπάρχει αντίστοιχο και πρόβλημα για τα κορίτσια, γιατί και εκείνα και τα... μιλάμε για κοινωνίες όπου οι γυναίκες είναι καταπιεσμένες. Ευχαριστώ. Ε, τον λόγο θα δώσω πρώτα στη Μαρτίνα για να απαντήσει για την κυδαιμονία. Ευχαριστώ. Μπορεί να είναι το πρόσωπο αυτό διοριζόμενο επίτημα, μπορούν δηλαδή να είναι από το συγγενικό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται άνθρωποι οι οποίοι ε, διαβιούν από μακρού στην ε, χώρα και βεβαίως ε, και, στο Βερολίνο υπάρχουν και πρωτοβουλίες που ε, προωθούσαν πρώην δικαστές, δικηγόρους και άλλους οι οποίοι αναλάμβαναν εθελοντικά. Η υποστήριξη δίνεται από τις αρχές προστασία του παιδιού υπό την επιτήρηση του δικαστηρίου. Υπό την εποπτεία του δικαστηρίου. Θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι, ορίστε. Εμείς έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς. Όταν αρχίσουν ε, τον επάγγελμά τους ε, περνούν από πρώτα, πρώτα από μία δεκαήμερη ε, ε, εκπαίδευση και μετά βέβαια στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν πολλές άλλες εκπαιδεύσεις. Τώρα, εμείς κάνουμε μια ε, αναθεώρηση του ε, δικαίου και έχω μια έκθεση για τα δικαιώματα των ασυνόδευτων παιδιών για να ενισχύσουμε τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται να διορίζεται κάποιος ως κυδεμόνας ή επίτροπος. Να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λευκοπινικό μητρό, να μην ε, έχουν ε, άλλα επιβαρυντικά στοιχεία κλπ. Τώρα, έχουμε στο άλλο ερώτημα εσείς Ευχαριστώ πολύ. Ορισμένα τμήματα του Αφγανιστάν θεωρούνται ασφαλή. Μπορεί να είναι ασφαλή, αλλά είναι στην περίπτωση αυτή σαν φυλακές. Εκεί υπάρχουν δε σημαντικές διακρίσεις. Δεν υπάρχει καμία χώρα που να εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση των φύλων. Στο κεντρικό Αφγανιστάν τα πράγματα είναι σχετικά ασφαλή, αλλά δεν μπορεί, για παράδειγμα, κανείς να ταξιδέψει σε άλλα τμήματα της χώρας. Δηλαδή είναι κανείς σαν κρατούμενος. Εφόσον ε, ταξιδέψει, κινδυνεύει να γίνει θέμα, ε, θύμα απαγωγής. Ορισμένες περιπτώσεις ε, δολοφονείται κιόλας, αποκεφαλίζεται και ούτω καθεξής. σε μια... Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη για δύο ε, ειδών λόγους. Το ταξίδι βέβαια είναι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα για τις γυναίκες είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετακίνηση αυτή. Στο δεύτερο βιβλίο μου έχω περιγράψει πως ένα 15χρονο κορίτσι προσπάθησε να διαφύγει. Όταν έφτασε στην Ελλάδα από το Αφγανιστάν είχε ήδη αποκτήσει δύο παιδιά από τους επαναλαμβανόμενους βιασμούς στη διάρκεια του ταξιδιού. Γι' αυτό και δεν τολμούν πολλά κορίτσια να ε, διαφύγουν, να ε, πάρουν το δρόμο της φυγής. Υπάρχει και το άλλο, το πολιτιστικό θέμα. Ο άνδρας είναι αυτός που φροντίζει για την οικογένεια. Οι τρομοκράτες άλλωστε τους άνδρες απευθύνονται και αυτούς προσπαθούν να στρατολογήσουν. Νεαρούς άνδρες. Ένας νέος ο οποίος απελάθηκε από την Νορβηγία το 2016 είδα φωτογραφίες του στην Συρία. Και ενώ ήταν χαρούμενος στην Νορβηγία, τον βλέπω τώρα πώς είναι στην Συρία μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι απελάβνονται δεν έχουν ε, πιθανότητα να επιβιώσουν. Είτε θα γίνουν εγκληματίες, είτε θα ε, προσχοληθούν στις δυνάμεις του Άσαντ ή από την άλλη πλευρά. Ευχαριστώ, Κατερίνα Κλίνιτς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους φιλοξενούμενους μας, μας για την ε, παρέμβασή τους ε, υπάρχουν διάφορες, ε, δια, ε, διάφορες υπάρχει μάλλον συγγνώμη, μια διακομματική ομάδα η οποία προσπαθεί να διαφυλάξει τα δικαιώματα των ανηλίκων και επειδή ούτως ή άλλως και εγώ επαγγελματικά προέρχομαι από, τον, από την προστασία των ανηλίκων, από το δικαστήριο ανηλίκων, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα και θα ήθελα απλώς να δείξω και κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ε, το μέγεθος του προβλήματος. Ο, αριθμός ε, των ε, ανηλίκων αυξάνεται, των ασυνοδεύτων ανηλίκων αυξάνεται και πολλοί ε, έχουν χάσει, ανήλικες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ταξίδι άφηξης. Είναι μια τραγωδία δηλαδή που μας θέτει ενώπιον των ευθυνών μας, σημαντικών ευθυνών και όπως ελέγχθη οι ανήλικοι μετανάστες ε, είναι παιδιά και για τα παιδιά είμαστε εμεί υπεύθυνοι και θα ήθελα να ρωτήσω α, ε, τους φιλοξενούμενους μας ε, να μου πούνε την ιδέα τους όσον αφορά την, την αλλαγή, της, την μεταρρύθμιση της διαδικασίας του Δουβλίνου κυρίως όσον τη χορήγηση του ασύλου, στο πρώτο σημείο εισόδου. Για τους, ε, μία, ε, για τους ασυνόδευτους ε, ανηλικούς αυτό αυξάνει την, τις πιθανότητες να αντιμετωπίσουν και περαιτέρω κινδύνους οι ανήλικες. Επίσης, η δυνατότητα χορήγησης βοήθειας και υποστήριξης, είτε είναι υγειονομική, είτε νομική, οτιδήποτε. Ε, δεν πρέπει να προσφέρουμε μόνο υποδοχή στους ανηλικές αλλά και ε, ε, υποστήριξη. Εδώ και λίγο καιρό στην Ιταλία έχουμε, έχουμε υπογράψει ένα πρωτόκολλο ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές, κυρίως στις τοπικές αρχές και στο το πρωτόκολλο αυτό υπάρχει ένας κατάλογος, ένα μητρό αν θέλετε, πιθανών κηδεμόνων. Στην Ιταλία ε, προσπαθούμε να Υπάρχει, μάλλον, ε, υπάρχει μια δυνατότητα στην Ιταλία να, να υποδεχόμαστε ή να υποδέχονται οικογένειες ε, τους ανήλικους μετανάστες. Λοιπόν, σε σχέση με την εμπειρία αυτή, έχουμε περίπου 2.000 παιδιά που ζουν σε φετές οικογένειες και πιστεύουμε ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και επιστημονική έρευνα γίνεται πάντα. Παρακολουθούμε τα παιδιά σε σχέση με την ανάπτυξή τους και αυτό που βλέπουν είναι ότι αν ζουν τα παιδιά σε θετική οικογένεια αναπτύσσονται καλύτερα. Κατά τα άλλα έχουμε κάποια μικρά κέντρα, τέσσερα παιδιά ε, ζουν μαζί, πρέπει να το σχάρει. Όσο μεγαλύτερες είναι οι δομές, όπως σας είπα, τόσο το χειρότερο. Βέβαια, το να θέτεις ε, τα παιδιά σε αυτές τις οικογένειες είναι κάτι πολύ καλό, στη δική τους πολιτισμό, στη δική τους κουλτούρα. Τα βοηθάει γιατί καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο για την κοινωνία, γιατί οι οικογένειες καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν για την ένταξή τους και πόσο δύσκολο είναι και υπάρχουν παραδείγματα πώς μπορούμε να το κάνουμε, αλλά ε, αυτό επειδή είναι οι άνθρωποι αυτοί από τις δικές σου ρίζες ε, βοηθά ουσιαστικά στην ένταξη, αλλά αυτό που χρειάζεσαι είναι επίτροπος, είναι ένας κηδεμόνας, γιατί θα πρέπει να υποστηρίξεις αυτές τις οικογένειες. Και μερικές φορές πρέπει να παρέμβεις, γιατί ενίοτε οι οικογένειες, ε, επειδή δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Μερικές φορές χρειάζονται βοήθεια, πρέπει να τους εξηγήσουμε τι να κάνουν, δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Ε, μερικές φορές ε, μπορεί να έχουν καλές προθέσεις, αλλά δεν λειτουργεί και πρέπει να είσαι επαγγελματία για να βλέπεις τι γίνεται, να έχεις ειδικές μεθοδολογίες, για να εξετάσεις τι γίνεται στις οικογένειες αυτές. Πρώτα είναι το θέμα της ασφάλειας. Αυτά τα προγράμματα έχουν ε, προκύψει από επιστημονική έρευνα. Έτσι λοιπόν αυτό πρέπει να εξετάζεται. Είναι πολύ καλό το σύστημα, αν υπάρχει επιτροπή, διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Τζακ Μάντισον, αντιπρόεδρο ε, της, ε, από την Εστονία, αντιπρόεδρο της Επιτροπής, μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στην Εστονία. Για τον κύριο Μαχμούντι. Έχω Εφόσον, εάν δούμε την Σουηδία, βλέπουμε ότι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών μελών η Σουηδία είναι από εκείνες που έχει υποδεχθεί πραγματικά πολλούς πρόσφυγες. Όμως, στα μίντια στη Σουηδία βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα. Φαίνεται πως προσέρχονται πολλοί στη Σουηδία, φτάνουν πολλοί στη Σουηδία. Πολλοί από αυτούς λένε ότι είναι λιγότερο από 18 ετών και καμιά φορά μετά αποδεικνύεται ότι είναι 25 χρονών και πάνω. Δεν είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι ανήλικοι. Είναι γνωστό ποιο ποσοστό από αυτούς ισχυρίζεται ότι είναι ανήλικοι και δεν είναι. Και μετά, εξετάζοντα τον χάρτη, πολλοί ε, πρόσφυγες ζητούν να πάνε μόνο στη Γερμανία, στη Σουηδία ή στη Φιλανδία, όχι σε άλλες χώρες. από το Τουρκμενιστάν για παράδειγμα. Δεν διεξάγεται πόλεμος εκεί. Γιατί έρχονται τόσο πολλοί στις ευρωπαϊκές χώρες και ζητούν να πάνε ε, οπωσδήποτε στη Σουηδία. Ενώ μπορούν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε άλλες χώρες ή σε χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο κοντά στο Αφγανιστάν και που δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει πόλεμο σε αυτές τις χώρες. Να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση πρώτα. 2,5 εκατομμύρια Αφγανοί πρόσφυγες ζουν στο Ιράν, περίπου 3 εκατομμύρια στο Πακιστάν. Πάρα πολύ μεγάλη αριθμή στο Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και αλλού. Εκεί όμως οι πρόσφυγες αυτοί δεν λαμβάνουν μόνιμη άδεια παραμονής. το Πακιστάν για παράδειγμα, που έχει 3 εκατομμύρια ε, Αφγανούς, απολάβνει, πολλού, απελάβνει, συγγνώμη, απελάβνει πολλούς από αυτούς. Τώρα, βεβαίως, όσοι επιθυμούν τώρα ε, να έρθουν στη Γερμανία, στη Σουηδία, μα αυτό ε, συμβαίνει διότι η Σουηδία προβάλλει μια καλή εικόνα ε, στο Αφγανιστάν. Ακούν οι Αφγανοί ότι η Σουηδία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα βέβαια μαθαίνουν σιγά σιγά ότι η ε, Σουηδία απελάβει όλο και περισσότερους, αλλάζει η εικόνα. Ήδη από το 2010-2011 μια μεγάλη ομάδα είχε ενσωματωθεί και από αυτούς άκουσαν μετά οι άλλοι που ήθελαν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς ε, που να πάνε. Άλλοι από αυτούς αποφάσισαν να ζήσουν, ε, να πάνε να ζήσουν στην Ουγγαρία και στην Ελλάδα, αλλά εκεί και από εκεί απελάβνονται. Τώρα για την πρώτη σας ερώτηση. Ούτε εκεί είναι απόλυτα σαφές ποια είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε συγκεκριμένες επιστημονικές αποδείξεις δεν μπορούμε να αποδείξουμε δηλαδή τη συγκεκριμένη ηλικία του ανθρώπινου όντως. Υπάρχουν κάποια τεστ, αλλά υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι επικρίνουν τα τεστ αυτά και θεωρούν ότι δεν μπορούν να δείξουν την πραγματική ηλικία. Και ούτε μπορεί κανείς να τη μαντέψει βεβαίως. Ε, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω ούτε και εγώ απάντηση στο ερώτημα σας αυτό. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα μιλήσω σου ειδικά. Α, όχι, όχι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ε, ένα λεπτό έχει ο καθένα ε, στην διάθεσή του πλέον. Κοιτάξτε. οι συναδελφοί μου θέσανε ερωτήσεις που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Στη Σουηδία το 2015 είχαμε 35.000 ε, ασυνόδευτους ανήλικους και είναι μικρή χώρα σχετικά. Δηλαδή το 40% όλων όσων ε, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 και 30 31000 ήταν νεαρά αγόρια. Ε, θέτω κάποιες ερωτήσεις δεν θα υπάρξει μια ανισορροπία, ε, δεν είναι ε, τελείως ε, δυσανάλογος ο αριθμός γυναικών και ανδρών, κοριτσιών και αγοριών, ένα κορίτσι για 11 αγόρια. Τέλο πάντων, είναι ένα θέμα που δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε, αλλά τέλο πάντων, μιλείς, είπατε ότι φύγατε από τον πόλεμο, φύγατε για να ξεφύγετε από τον πόλεμο. Πώς μπορείτε να, πώς τι, πώς γίνεται να περάσετε από όλες αυτές τις χώρες ε, και να φτάσετε από όλες αυτές τις χώρες ε, και να φτάσετε στη Βόρεια Ευρώπη. Γιατί δεν πήγατε ας πούμε στην Δανία, στην Φιλανδία ή στην Νορβηγία και ήρθατε στη Σουηδία. Τι έχει η Σουηδία. Απήντησα ήδη ότι πάρα πολλοί άνθρωποι φεύγουν γιατί θέλουν να αποφύγουν τον κίνδυνο. Θέλουν να αισθάνονται ασφαλείς και στις χώρες του Νότου, από τις χώρες του Νότου μάλλον, θα απελαθούν κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα. Άρα ψάχνουν να βρουν μια ασφαλή χώρα και η, η Σουηδία θεωρείται ασφαλής. Από την άλλη πλευρά δεν είναι και πάρα πολλοί που μπορούν να μπουν στην, στη Σουηδία. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή τη δυσαναλογία ανάμεσα στον αριθμό αγοριών ή και κοριτσιών. Τι γίνεται με τα κορίτσια. Εάν ένα, μια γυναίκα, μια νεαρή κοπέλα βγει μόνη της στο δρόμο, έχει, αντιμετωπίζει προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Αν όμως έρθει στην Ευρώπη ε, θεωρείται, αν θέλει να έρθει να πάει στην Ευρώπη, θεωρείται ότι ε, ε, παραβιάζονται οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας και μπορεί να φτάσουμε και μέχρι λιθοβολισμό, όταν, αν πάει να κυκλοφορήσει και μόνο τη στον δρόμο. Άρα, τέλος πάντων, είναι θέμα νοοτροπίας της κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της Επιτροπίας που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το θέμα του σχολείου, της εκπαίδευσης. Μιλήσαμε πάρα πολύ για τους συνοδευτούς ενηλίκους, αλλά πρέπει να ακούσουμε και από εσά τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό με ενδιέφερε εμένα. Ε, και εγώ είμαι Σουηδή και είμαι περήφανη για το γεγονό ότι τόσοι άνθρωποι φτάνουν στη Σουηδία γιατί έχουμε μια χώρα ισότητας ε, και βέβαια ακόμη πολλά πρέπει να γίνουν αλλά προσπαθούμε να μεταχειριστούμε σωστά τους ανηλίκους και να περάσω στο επόμενο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν ε, πρέπει να μεταχειριζόμαστε διαφορετικά τους ανηλίκους οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, ακόμη και αυτοί που έρχονται και με τους γονείς τους, θα πρέπει να χαίρουν τις ίδιες μεταχείρισης. Δεν πρέπει να ζημιώνουμε τους ανθρώπους αυτούς. Και άκουσα τι είπε ο Μιντ αν ε, δεν σκεφτούμε να τους δώσουμε μόνιμη άδεια παραμονής, δεν μπορούν διαφορετικά να έχουν ασφάλεια οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστώ. Λέει ο κ. Λόπες Αγγιλάρ. Νομίζω ότι ήταν ε, η πιο ενδιαφέρουσα συνεδρίαση σήμερα. Φυσικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η μαρτυρία του κ. Μαχμούντι. Όμως, Θέλω να σας ε, ρωτήσω κάτι, κύριε Φερστέγγεν. Καθώς ε, δώσατε ιδιαίτερη προσοχή στο ποια είναι, ε, ο, ποιος είναι ο τρόπος προσέγγισης ενός ενηλίκου από την Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Είπατε ότι πάρα πολλά παιδιά ήταν θύματα εμπορίας, ανθρώπων, εκμετάλλευσης κτλ. Ακούσαμε ότι η έκθεση, ότι η Europol ανέφερε ότι 10.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι αγνοούνται. Και πώς εξηγείται ότι μπαίνουν σε αυτό το κύκλωμα εκμετάλλευσης οι ανήλικοι και πώς μπορείτε εσείς, πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό. Κοιτάξτε, στις κατοχώρες ε, δεν είναι ότι μπορούμε να το προλάβουμε, αλλά έχουμε κάνει πολλά. Και σας είπα ότι έχουμε χώρους προστασίας, καταφύγια, Παραδείγματο χάρη για τα κορίτσια από την Ιγυρία όλα αυτά τα κορίτσια εξαφανίστηκαν πριν και στο τέλος του project το 85% εξακολουθούν να βρίσκονται στις κάτω και συλλάβομαι 69 ε, διακινητές όχι μόνο στις κάτω αλλά σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται λοιπόν για συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων. Αν συνεργαστούν όλοι αυτοί δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά όχι μόνο στις κατοχώρες, πρέπει και διασυνοριακά τότε μπορείς να κάνεις κάτι. Αλλά καθημερινά πρέπει να διδασκόμαστε. Δεν τους χάρη για τα παιδιά από το Βιετνάμ που έρχονται τώρα στις κατοχώρες και αυτά αγνοούνται και δεν κατανοούμε γιατί εξαφανίζονται τα γόρια από το Βιετνάμ. Την επόμενη φορά που θα είμαι εδώ θα σας εξηγήσω γιατί και πώς θα το σταματήσουμε. Γιατί αυτό πρέπει να σκεφτεί κανείς. Δεν μιλάμε για μία και μόνη λύση. Και αν ε, Θέλετε, θα ήθελα να απαντήσω και στο γιατί επιλέγουν τη Σουηδία. Έχει συμβεί και στις κατοχώρες. Το 2001 είχαμε το ίδιο πρόβλημα γιατί όλοι αποφάσισαν να πάνε στην Ολλανδία και οι πολιτικοί έλεγαν ε, τότε ότι επειδή τον ίδιο θα πάει πολύ καλά. Και γι' αυτό άρχισαν να κάνουν κάτι διαφορετικό επειδή ήταν ε, πάρα πολύ κατά πράγματα στις κατοχώρες. Αν ρωτήσετε τώρα τα παιδιά γιατί πάνε στις κατοχώρες στη Σουηδία, θα έχετε την ίδια απάντηση που είχατε και πριν. Δεν κάναμε την επιλογή, άλλοι έκαναν την επιλογή και ε, μερικές φορές ζει σε μία φούσκα για δύο χρόνια. Τόσο διαρκεί το ταξίδι σου και απλώς συναντάς ανθρώπους που είναι σε φυγή και απλώ ε, γνωρίζει διακινητέ και όλοι σου λένε μια ιστορία. Και είναι η ίδια ιστορία γιατί είναι μέσα σε αυτή τη φούσκα. Αν θες να το σταματήσεις αυτό, πρέπει ε, τελικά να ξεκινήσεις ε, ε, από όταν μπαίνουν τα παιδιά αυτά στην Ευρώπη. Να υπάρχει ο επίτροπος από τη στιγμή που μπαίνουν, να το ενημερώσει το παιδί ποιον μπορεί να εμπιστευτεί και τότε μπορεί να γίνει ε, μια κατάσταση που να αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο αυτό. Όμως, σας παρακαλώ, μην μειώνετε την φροντίδα δεν ε, διαλέγουν λόγω της καλής φροντίδας, απλώς ε, ψάχνουν κάποιες ευκαιρίες για το μέλλον τους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα με την κυρία Ροντρίγες από την Ισπανία. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τους ομιλητές στο πάνελ, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε. Δύο ερωτήσεις. Θα ήθελα την άποψή σας για το εξή. Για το αν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μπορούν να, να τεθούν υποδικητική κράτηση όσο εξετάζεται το αίτημά του. Η θέση τη είπα τη αρμοστία ήταν σαφή ότι σε καμία περίπτωση κανένα ενήλικο δεν μπορεί να τεθεί υποκράτηση επειδή έχει μπει παράνομα σε μια χώρα ή είναι παράνομο. Και η βάση και τη ε, σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού ποτέ δεν επιτρέπεται η κράτηση γιατί θίγει τα συμφέροντα του παιδιού. Θέλω να ρωτήσω και κάτι τον εκπρόσωπο της Νίντο. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, πώς το επιλύετε. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας ε, ανήλικος, ο οποίος είχε επίτροπο και ενηλικιωθεί, τότε τι υπερισχύει ε, υπερισχύει ο νόμος περί αλλοδαπών ε, ή η κατάστασή του ε, ότι χρήζει προστασίας. Γιατί είχαμε μία ανώμαλη κατάσταση εμείς, παραδείγματος χάρη, είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε ζητήσει άδεια παραμονής, γιατί έχριζε προστασία ως ενήλικος και τελικά μετά τα 18 μπορεί να βρεθεί στο δρόμο. Τώρα στην Ισπανική νομοθεσία αναφερόμαστε στους ε, ανθρώπους που δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η ηλικία τους. Στο άρθρο 49 της Ισπανικής νομοθεσίας λένε ότι αμέσως ουσιαστικά χρήζει προστασία. αν υπάρχουν αμφιβολίες γίνονται κάποια τεστ. Αλλά ε, αν υπάρχει άρνηση από ε, τον άνθρωπο να κάνει αυτά τα τεστ, παρόλα αυτά διαβιβάζεται η αίτησή του στην αρμόδια εισαγγελία. Ευχαριστώ κυρία Γκρισβέκ. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα με λίγα λόγια και εγώ να χαιρετήσω την ποιότητα, την δύναμη και την λογική όσων πήραν το λόγο σήμερα το απόγευμα ε, πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό για τα παιδιά τα ίδια αλλά και για το αυτό ε, που αντιπροσωπεύει η Ευρώπη όταν υποδέχεται ασυνόδευτους ανήλικους θα απλουστεύσω την ερώτησή μου, μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ούτως ή άλλως τα περισσότερα θέματα εθήθηκαν τα πιο σημαντικά. Ε, η αξιολόγηση της ηλικία, ε, η φιλοξενία των ε, παιδιών, το θέμα του κηδεμόνα, όλα αυτά τα θέματα αποτέλεσαν και αντικείμενα ανάλυσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ξαναστείλω την μπάλα, αν θέλετε, το μπαλάκι στο δικό σας κομμάτι του γηπέδου, μια και μιλάμε για το άσυλο. Ε, υπάρχουν διάφορες διατάξεις για τα ευαίσθητα άτομα, μεταξύ αυτών και τα παιδιά βέβαια. Λοιπόν, θα ήθελα να ξέρω τις προτάσεις σας όσον αφορά και τις απόψεις όσον αφορά το, το άσυλο, το πακέτο αυτό για το άσυλο. Ε, Ποιε είναι οι προτεραιότητε, σα, παραδείγματος χάρη, γιατί υπάρχουν διάφορες διατάξεις ε, τις οποίες εξετάζουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, μια διάταξη που είναι αντίθετη με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε ένα παιδί από, το ένα, από τη μία χώρα στην άλλη έτσι σαν πακέτο. Ε, εγώ θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες σε σχέση με το κείμενο το οποίο προσπαθούμε να συντάξουμε, να οικοδομήσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Η Πάολα Μπίλερ από την Σουηδία. μια και άκουσα τον Μαχμούντι κατά τη διάρκεια του γεύματο, είχα την τύχη να κάθομαι δίπλα του, ε, θα ήθελα να θέσω τι ερωτήσεις μου στους άλλους δύο, για τις κοπέλες ε, που είναι παντρεμένε. Χρειάζονται, επειδή υπάρχει νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ηλικία ε, γάμου Ε, παιδιά, κορίτσια τα οποία παντρεύονται σε ηλικία 16-17 ετών ε, χρειάζονται ειδικό πιστοποιητικό για να παντρευτούν και γιατί κάνετε διάκριση ανάμεσα ε, στα κορίτσια που προέρχονται από τη χώρα σας και κορίτσια τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες. Μιλήσαμε λίγο για τα τεστ τα οποία είναι διαθέσιμα ε, για τα, γίνονται τα τέστα αυτά και στην χώρα σας ε, ε, αρχιά, στην αρχή της διαδικασίας και αυτά τα τέστα μπορεί να γίνουν και στη Σουηδία για να δούμε τα παιδιά αυτά, τα κορίτσια αυτά είναι ανήλικα. Επίσης, δυστυχώς στην Σουηδοί δεν έχουμε πολλές ε, ε, οικογένειες ε, που υιοθετούν παιδιά ή φιλοξενούν παιδιά. Ζουν σε κέντρα. Έχετε διαφορετικά κέντρα για τους εφήβους, παραδείγματος χάρη στη δική σας χώρα. Ή εάν είστε σίγουροι ότι πρόκειται για παιδιά, υπάρχει ένα διαφορετικό ε, έντες χώρο χώρος φιλοξενίας. Και εγώ είχα την χαρά να μιλήσω με τον κύριο Μαχμούδη όταν επισκεφθήκαμε την Σουηδία και μάλιστα μετά από μια καταθλιπτική ημέρα όπου η Σουηδική αστυνομία μας είχε πει ότι δεν έχει αρκετούς ερευνητές για να ψάξουν να βρουν τους ασυνόδευτους ανηλίκους που είχαν εξαφανιστεί. Και λέω προ τιμή τη ειδική αστυνομία ήταν πολύ αναστατωμένη για το λόγο αυτό. Και είδαμε μετά τον κύριο Μαχμούδη και του φίλου του, και ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα. Και είναι πολύ σημαντικά τα όσα μα είπατε. Και ιδίω να διαλυθεί ο μύθο ότι δίθεν το Αφγανιστάν είναι ασφαλή χώρα. Δεν είναι. Δεν είναι ασφαλής χώρα το, το Αφγανιστάν. Και εσεί, κύριε Παστάκεν χρειάζεται πρόγραμμα να αντιμετωπίζονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στι χώρε όπου εισέρχονται στην Ευρώπη και όπου αντιμετωπίζουν του κινδύνου και όπου πολλοί από αυτούς όπως οι Αφγανοί τους αρνούνται την είσοδο διότι δεν ε, εκπληρούν τα κριτήρια. Το ε, αντίθετο πρόβλημα έχουμε εμεί στην Πορτογαλία από τη Σουηδία. Εμεί θέλουμε πρόσφυγε και μάλιστα θέλουμε και ανήλικου για να αντιμετωπίσουν και τα, όλα του τα προβλήματα. Που θεωρούμε ότι οι περισσότεροι από αυτού του ανηλίκου, ε, Αφγανοί, ε, παιδιά από το Αφγανιστάν, που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, για παράδειγμα στην Ελλάδα. Και δεν έχουμε το νομικό πλαίσιο για να τους δοθούν αυτές, να τους δοθεί αυτή η προτεραιότητα σε αυτούς τους νέους αυτούς ανηλίκους που έχουν τη μεγάλη ανάγκη προστασίας. Ευχαριστώ, Άννα. Μαρτίνα. Αρχίζει τώρα και ζεσταίνεται η συζήτηση και κρίμα που είναι προχωρημένη ώρα, γιατί δεν μπορώ βέβαια να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα, γιατί δεν προλαβαίνω, αλλά κάθε άνθρωπος αναζητεί μια ασφαλή προοπτική και πιο πολύ από όλα τα παιδιά αυτά. Η ιδέα ασφαλής προοπτική θα πρέπει να δοθεί το δυνατόν συντομότερο. Από την άποψη του δικαίου αλλοδαπών όμως χρειάζεται χρόνος και ειδικά για την περίοδο αυτή πρέπει να εξηγείται με αλφαγιώτα δηλαδή στα παιδιά ποια πράγματα απαιτούνται και να τους δημιουργείται εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντική αυτή η επιτροπή, η κυδαιμονία. Όταν τα παιδιά αυτά ενηλικιώνονται μετά υπάρχει ένα σύστημα χορήγησης βοήθειας σε νεαρούς ενηλίκους πλέον. Και αυτό τους εξηγείται και ε, συνοδεύονται στα διάφορα βήματα ώστε να μπορέσουν να περάσουν μετά σε αυτό το σύστημα. Σύμφωνα με το εθνικό μας δίκαιο στη Γερμανία πάντα από 16 ετών και άδνο βρίσκεται το άτομο στην νόμιμη ηλικία γάμου, Εφόσον όμως το δεχτεί το δικαστήριο. Το δικαστήριο όμως όλο και λιγότερο δέχεται την υπόθεση αυτή, διότι δεν ταιριάζει με τις απόψεις της κοινωνίας. Και όπως σας εξήγησα υπάρχουν κάποιες τροποποίησεις του νομοσχεδίου και ε, θα πάψουν να δίνονται οι άδειε αυτές και η νόμιμη ηλικία γάμου θα είναι από τα 18 και μετά. Verstegen, να αρχίσω με την ηλικία μετά τον τα 18 και να σας πω μετά και για την Επιτροπή η Κυδαιμονία. Είναι το πρόβλημα αυτό βέβαια μετά από τα 18. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Για τους δικαστές είναι πρόβλημα. Η τοποθέτηση σε ανάδοχες οικογένειες βοηθάει, διότι οι οικογένειες αυτές δεν τους ξαποστέλουν και μετά τα 18, εάν μείνει στην Ολλανδία, σημαίνει ότι μπορεί να πα στο σχολείο. Να βρει δουλειά. Αρχίζουν ήδη από τα 17, όμω, διότι πρέπει να του προετοιμάσει κανεί για τα 18. Όμω τοποθετούνται σε ανάδοχε οικογένειε, ή σε μικρέ μονάδε ένα σπίτι για μια οικογένεια, σε μικρού δρόμου και φορά μπορεί να μείνουν τα παιδιά αυτά εκεί, μένουν στην τοπική κοινότητα η οποία είναι υπεύθυνη για αυτούς. Έτσι λοιπόν ε, κάνουμε συμβάσεις με αυτούς. Θα, λέμε θα τοποθετήσουμε τα παιδιά στην κοινότητά σας αλλά θα πρέπει να τους βρείτε στέγη μετά από τα 18 τους χρόνια και να τους δώσετε και κάποια ε, κατεύθυνση, κάποια guidance είτε με κοινωνικούς λειτουργούς ή με άλλο τρόπο. Αυτά για να σας δώσω μια σύντομη εξήγηση. όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών τοποθετούνται σε ανάδοχε οικογένειε, διότι όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών είναι ευάλωτα. Αυτό λοιπόν γίνεται από την πρώτη στιγμή που φτάνουν στην ε, Ολλανδία. Για την εκτίμηση τη ηλικία. Έχουμε ένα σύστημα εκτίμηση ηλικία ε, και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει τέτοιο σύστημα. Κάνουμε ακτινογραφίες των καρπών καθώς και του οστού ε, στον ε, θώρακα που σας δείχνανε 18 και άνω. Αν όμως δεν έχει κλείσει το οστό αυτό, τότε είστε μεταξύ 16 και 32 ετών. Ε, υπάρχει βέβαια πάντοτε το ευεργέτημα της αμφιβολίας αν δεν έχει κλείσει το οστό αυτό στο κέντρο του θώρακος. Έχουμε λοιπόν την εκτίμηση Όταν αρχίσαμε, θεωρούσαμε ότι πάνω από τα, βρήκαμε ότι πάνω από τα 50% αυτών που έλεγα ότι είναι κάτω των 18 ετών ήταν στην πραγματικότητα πάνω από 23. Δεν το χρησιμοποιούμε πλέον το σύστημα αυτό, δεν το, δεν το χρειαζόμασταν, αλλά τώρα όμως θα ξαναρχίζει η προσέλευση μεγάλων αριθμών που σχίζει την 118 και θα ξαναρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Έτσι λοιπόν Βεβαίω η ακτινογραφία είναι δύσκολο να ληφθεί με τον ορθό τρόπο κλπ. Δεν είναι η απόλυτη λύση, αλλά βοηθάει πολύ. Τώρα για το Δουβλίνο, ναι, να πω. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι κατά τη γνώμη μας δεν μπορείτε να αποκτήσετε κηδεμόνα στην χώρα που βρίσκεστε αν δεν τον έχετε από την πρώτη χώρα. θα πρέπει να περάσετε από ένα κηδεμόνα σε άλλον, έρθει δηλαδή ο δεύτερος σε επαφή με τον πρώτο για να γίνει σωστά. Και τότε θα φανεί αν είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Και το παιδί καταρχήν θέλουμε να μπορεί να διαμένει στους κόρπους μιας οικογένειας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Τέλος, τα παιδιά που διαμένουν σε άγνωστη διαμονή. Έχουμε ένα ποσοστό 15% τα οποία ε, φεύγουν, παλαιότερα ήταν 15%, ε, φεύγουν με άγνωστο προορισμό. Τώρα έχουμε φτάσει στο 5%. Από τις οικογένειες δεν εξαφανίζονται. Από μικρές μονάδες μάλλον δεν φεύγουν. Μετά είναι και βέβαια και τα κέντρα υποδοχής. Από εκεί πράγματι εξαφανίζονται. όσο πιο στενός είναι ο σύνδεσμος με τον κηδεμόνα, τόσο περισσότερο τείνουν να παραμένουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και του συναδέλφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια για αυτή την ιδιαίτερα καρποφόρα συζήτηση. Έμαθα πάρα πολύ, ήταν εξαιρετικό το πάνελ και θα ήθελα να του χειροκροτήσουμε. And please, let's continue. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Έχουμε τώρα το πακέτο ασύλου και ευρωπαϊκούς κανόνες. Ο λόγος που τα τροποποιούμε είναι επειδή δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και είναι σημαντικό να συνεργαστούμε για να δυσφαλίσουμε ότι λειτουργεί η ελληνική στην πραγματικότητα και ότι όλα τα κράτη-μέλη επιμερίζονται την ευθύνη στο να θέσουμε στο επίκεντρο το συμφέρον του παιδιού και να εξυπηρετήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα τα συμφέροντα του παιδιού. Ευχαριστώ πολύ. So, colleagues, um, I think we are now going to... Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε στην καταληκτική συνεδρίαση. Ξέρω ότι κουραστήκατε γιατί ήταν ε, μακρά ημέρα, αλλά όσοι μπορείτε να παραμείνετε θα έχουμε μια σύντομη καταληκτική συνεδρίαση.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 Okay, dear colleagues, um... Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι ορισμένοι φεύγετε και αντελάστε κάρτες και τα λοιπά, πολύ ωραία, αλλά για όσους μείνετε να περάσουμε στην καταληκτική συνεδρία, μπορείτε να αποχαιρετιστείτε κάπου αλλού. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Από καταλαβαίνω είναι πολύ λίγοι άνθρωποι εδώ, αλλά θα ήθελα καταρχήν να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη των κοινοβουλίων. Ξέρω ότι κάποιοι έπρεπε να αποχωρήσουν. Ευχαριστώ και όσους παραμένουν. Ευχαριστώ και το προσωπικό τους. Έχουμε... Εντάξει, το δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που έμειναν σε όλη τη συνεδρίαση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να διασφαλίσουμε ότι οι δέσμοι μέτρων για το άσυλο θα συζητηθεί και ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν και στα εργαστήρια και φυσικά και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που ήρθαν από μακριά. Δεν θα κάνω τώρα κάποιες ε, τελικές παρατηρήσεις, ε, θα περάσουμε στις συστάσεις των εργαστηρίων. Όμως δεν θέλω να μακρηγορήσουμε γιατί έχουμε και μία παρουσίαση. από την πρωτοβουλία ένταξη του ποδοσφαιρικού ομίλου του Κράινε. Θέλουμε να τους ακούσουμε και αυτούς τους καλέσαμε να έρθουν ε, από κάπως μακριά. Θέλουμε να τους ακούσουμε. Θα, προσ... θα έχετε προσέξει ότι πρέπει να έχουμε εδώ συστάσεις των εργαστηρίων. Ε, δύο από τους πρόεδρους δεν μπορούν να είναι εδώ. Μία από τους πρόεδρους παρέμεινε, Κορνίλια. Αυτό είναι επειδή είσαι καταπληκτική. Σε ευχαριστώ που έμεινες. Και καθώς ε, επανήλθες, Κορνήλια, θα ήθελα να σου ζητήσω να μας κάνεις και μία σύντομη ενημέρωση. Αν συμφωνείς, θέλω να προτείνω το εξής. Δεδομένου ότι και πολλά μέλη της ΛΥΜΠΕ έπρεπε να αποχωρήσουν, θα ζητήσω από την κυρία Ένστε να κάνει την, την παρουσίασή της. Ε, οι άλλοι δύο πρόεδροι έδωσαν κάτι γραπτός. Και αυτό που θα ζητήσω είναι καταρχήν να πάρει το λόγο η κυρία Έρνστ και κατόπιν εγώ θα παρουσιάσω μια πλήρη αναφορά από όλα τα εργαστήρια που θα μοιραστεί και σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου συντομότατα όταν ολοκληρωθεί αυτή η συνεδρίαση και στα μέλη της ΛΥΜΠΕΡ. Θα πρέπει κύριε Σιμπλ κύριε Μπέκερ να παρουσιάσουν με δικά τους λόγια τα εργαστήρια. Δεν νομίζω ότι δεν είναι καλό να τα διαβάσω εγώ. Παρακαλώ, Κορνίλια, έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομη. Ήταν πολύ σημαντικό το θέμα της σημερινής διαταξή διαταξής μας, δηλαδή τα δικαιώματα των θυμάτων του, της εμπορίας ανθρώπων. Είχαμε και την κυρία Σεκελιάδου, εκπρόσωπο της κυρίας Βασιλιάδου, μέσα σε ένα χρόνο 16.000 θύματα του εμπορίου αυτού. 65% των θυμάτων είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι προκαλείται το εμπόριο αυτό ανθρώπων μόνο από τα μεταναστευτικά ρεύματα και ρεύματα προσφύγων. Μιλήσαμε για την σεξουαλική εκμετάλλευση, για την εκμετάλλευση της εργασίας των προσώπων αυτών σε διάφορους τομείς καθώς και για άλλα πράγματα όπως εμπόριο οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Εκεί έχουμε πάρα πολύ λίγα στοιχεία βεβαίως. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι συλλέγονται δεδομένα στις χώρες μέλη, αλλά ε, για να γίνει αυτό πρέπει να γνωρίζει κανείς τι σημαίνει ότι κάποιος είναι θύμα του ε, εμπορίου ανθρώπων θα πρέπει και οι αρμόδιες αρχές να είναι ενήμερες και εκπαιδευμένες, αλλιώς δεν μπορούν να εντοπιστούν τα θύματα αυτά, ούτε να ληφθούν μέτρα. Λοιπόν, αυτή η ενημέρωση και η εκπαίδευση δεν είναι αρκετά προχωρημένη στις διάφορες χώρες μέλη. Χρειάζεται λοιπόν να εξεταστεί στο σοβαρά το θέμα αυτό, να βρεθούν ποια είναι τα θύματα αυτά για να τους χορηγεί βοήθεια. διαμορφώνεται τώρα το πλαίσιο για να διασφαλίζονται καλύτερα τα δικαιώματα των θυμάτων του εμπορίου ανθρώπων και είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς ότι αυτό δεν ωφελεί, το εμπόριο αυτό ωφελεί πολλούς, τους παρόχους υπηρεσιών, ορισμένους κλάδους της οικονομίας, όχι μονάχα δηλαδή τους ε, παρανομους διακινητές. Αν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η μαύρη αγορά δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Ως συμπέρασμα τώρα, μετά από μια πολύ ζωηρή συζήτηση, το συμπέρασμά μας λοιπόν ήταν το εξή. Πρώτον, εντείνεται το εμπόριο παιδιών. Αυτό το ζήτημα πρέπει να περάσει σε όλα τα νομοθετήματα που έχουν σχέση με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Για παράδειγμα, παράνομες υιοθεσίες ε, εμπόριο οργάνων, ανθρώπινων οργάνων, να, πρέπει να μιλήσουμε και για τα αγνοούμενα παιδιά. Ένα ανοιχτό πρόβλημα, όπως γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό να τα σημειώσουμε όλα αυτά. Εμπόριο παιδιών, ξαναλέω, εκμετάλλευση παιδιών αλλά και γυναικών. Δεν υπάρχει καμιά χώρα μέλος που να μην σημειώνεται εμπόριο ανθρώπινων όντων. Καμία δεν βρίσκεται στο πράσινο, το πω έτσι ακόμα και για χώρες που δεν το περιμέναμε, ακούσαμε τα πράγματα αυτά. Και όλες οι χώρες μέλη πρέπει να επαναξετάσουν τις νομοθεσίες τους και να φροντίσουν να εφαρμοστεί η οδηγία. Η αποζημίωση των θυμάτων στις περισσότερες χώρες δεν λαμβάνει χώρα. Είναι όμως ένα σημαντικό θέμα το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να ρυθμιστεί. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει ε, ποινική δίωξη των θυμάτων, γιατί για παράδειγμα πέρασαν παράνομα τα σύνορα, βεβαίως εφόσον τους διακίνησαν οι παράνομοι διακινητές και ούτω καθεξής. Πολύ σημαντικό επίσης, όταν δηλαδή τα πρόσωπα αυτά είναι θύματα ε, τέτοιων εγκλημάτων, πρέπει να μπορούν να κλητεύονται και ως μάρτυρες. Πρέπει να προστατευτούν και τα δικαιώματα των μελών της οικογένειας. Υπάρχει συχνά το στίγμα. Αν όλα αυτά δεν τα αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. συζητούμε, συζητήσαμε μάλλον και για ενδεχόμενες προσφυγές επί παραβιάση, γιατί πολλές ε, χώρες μέλη διαφορούν για την εφαρμογή της οδηγίας. Όπως είπα και πριν, πρέπει να είναι δυνατόν να εντοπίζονται τα θύματα. Αυτό χρειάζεται κατεπηγόντως εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε όλες τις χώρες μέλη όλων των ε, ε, αξιωματούχων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. σε περίπτωση ε, λαθρέας διακίνησης ανθρώπων. Είναι διαφορετική, για παράδειγμα, υπόθεση από την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Το μέρα θέμα, όπως είπα, είναι η διακίνηση των παιδιών. Για όλες τις οδηγίες πρέπει να μπει το θέμα, να μπουν τα θέματα αυτά να ρυθμιστούν σε όλες τις οδηγίες, γιατί αλλιώς όλες οι προσπάθειες που κάνουμε είναι εισμάτιν. Ευχαριστώ Κορνέλια. Ευχαριστώ. Έτσι όπως είπαμε και σε άλλα παράλληλα εργαστήρια, ούτως ή άλλως θα έχουμε μια γραπτή έκθεση η οποία θα υποβληθεί σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ε, ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στις ε, συνεδρία, στις συναντήσεις. Βέβαια χάνουμε, φιλορροούμε όσο περνάει η συζήτηση. Ε, ας ακούσουμε τώρα από τους φίλους μας, από την ποδοσφαιρική ομάδα που ζητάνε για κάτι θετικό. Πολλοί συνάδελφοι με ρωτήσαν γιατί να μην ε, κάνουμε και κάτι θετικό όσον αφορά ε, την χορηγησία ασύλου και τους ανήλικους. Ε, υπάρχει και το γεγονός ότι πρέπει να συζητήσουμε και τα θέματα αυτά και με τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, και είναι καλό να έχουμε εδώ και εκπροσώπους των προσφύγων και των μεταναστών. Έχουμε δύο Έχουμε εδώ εκπροσώπους από την ε, ποδοσφαιρική ομάδα του Κράινεμ ε, που θα παρουσιάσουν την ε, πρωτοβουλία τους. Ο Νίο Κίνε και ο Μπέντζαμιν Ρενό είναι θελοντές, ενώ ο Τιερί Πία και ο Γκρέγκορι Μπλακ είναι οι διευθυντές του κέντρου Φενταζίλ που είναι οι τοπικές αντένες, αν θέλετε, της ε, Βελγικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την υποδοχή των ετούντων άσυλων. Ε, δεν Νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο για να ακούσουμε όλους. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ ε, και θέλει να μας παρουσιάσετε τα θετικά, ένα θετικό παράδειγμα για την ένταξη των τον άσυλο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Προτείνω να ξεκινήσουμε με το βίντεο για να καταλάβετε ποιο είναι το project μας. Je je m'appelle Gabriel, j'ai 10 suis de et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 Uh, Καλησπέρα σε όλους. Ίσως μπορούμε να συνεχίσουμε μια παρουσίαση PowerPoint. Ε, είδατε ότι αυτό το βίντεο έγινε από ε, το Ίδρυμα του Βασιλιά Μποντουά. Να κάνω μια σύντομη παρουσίαση του κλαμπ μας. Καταρχήν, ε, είμαστε ένα σύλλογος στο Κράινεμ, έξω από τις Βρυξέλλες. Αυτή είναι τώρα η ιδιαιτερότητα, είναι η πολυπολιτισμικότητα, όχι μόνο έχουμε 300 παίκτες, αλλά προέρχονται και από 40 διαφορετικές χώρες. Έτσι λοιπόν, ε, βλέπετε εδώ ότι αναμειγνύονται διάφορες κουλτούρες και διάφορα κοινωνικά background. Αυτό μπορεί να το κάνει το ποδόσφαιρο. Φέρνει μαζί ανθρώπους από διαφορετικά background που διαφορετικά δεν θα γνώριζαν στον άλλο. Και Ακριβώς εδώ θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτό το project. Το ξεκίνησαμε το Σεπτέμβριο του 2015. Είναι το δεύτερο έτος τώρα που διανύουμε. Η ιδέα μας ήταν ως ε, ένα πολυπολιτισμικός ε, ποδοσφαιρικός ε, σύλλογος να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα για την ένταξη των προσφύγων. Σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Φεντασίλ και να έρθουν οι πρόσφυγες ε, στον ομιλό μας να παρακολουθήσουν και μάθημα γαλλικών και να κάνουν ε, και μια εκπαίδευση στο ποδόσφαιρο. Είχαμε 700 ε, πρόσφυγες την πρώτη περίοδο και τώρα συνεχίζουμε στην διαβάση με τη δεύτερη περίοδο. Έχουμε καθημερινά 6 με 10 πρόσφυγες, τρεις φορές την εβδομάδα έρχονται. Έτσι λοιπόν, καταρχήν έχουμε το μάθημα γαλλικών ο Άλμπο που είναι καθηγητής, θα μιλήσει γι' αυτό αργότερα. Αυτό ήταν ε, πολύ σημαντικό για μας, ε, γιατί ουσιαστικά θέλαμε να τους δώσουμε για κάποιες έννοιες της γλώσσας. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντάξεις ανθρώπους ε, στη χώρα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ έχουμε την κατάρτιση στο ποδόσφαιρο, βλέπετε και στην φωτογραφία, προσπαθούμε να τους ε, αναμίξουμε με τους δικούς μας παίκτες. Δεν θέλουμε να έχουμε ξεχωριστή εκπαίδευση, ξεχωριστή προπόνηση, αλλά θέλουμε να τους εμπλέξουμε στις ε, ομάδες νέους. Έχουμε μικρές ομάδες, τρεις-τέσσερις παίκτες και τους βάζουμε σε μια ομάδα με ανθρώπους ίδιας ηλικίας, συνομιλίκους τους είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επαφή μεταξύ προσφύγων ε, και ε, των δικών μας παικτών, γιατί διαφορετικά δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, ξέρετε, είναι πιο εύκολο να είσαι με τους δικούς σου φίλους, επειδή μιλάτε την ίδια γλώσσα. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε να τους βγάλουμε από αυτή την άβολη κατάσταση. Στην επόμενη διαφάνεια Βλέπετε μια πολύ σημαντική πτυχή. Εδώ έχουμε κάθε βράδυ μετά την προπόνηση ένα δείπνο όπου τρώνε όλοι μαζί και αυτή είναι η στιγμή που γνωρίζεις τους ανθρώπους αυτούς, τους μιλάς, μπορεί να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, ακούς τις ιστορίες τους, τι έχουν περάσει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα, δεν πρέπει να το εκοτιμούμε. Μελλοντική στόχη δεν ε, θέλουμε να γίνει κάτι άπαξ, θα κάνουμε και μια τρίτη εποχή την επόμενη περίοδο και γιατί να μην συνεχίσουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο συλλόγων στο Βέλγιο αλλά και στην Ευρώπη και να έχουν το ίδιο όραμα που έχουμε και εμείς. Θέλουμε να εξάγουμε το project μας και σε άλλους συλλόγους, να τους πείσουμε να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες. Συνεργαζόμαστε και με την Ποδοσφαιρική Ένωση του Βελγίου και προσπαθούμε να πείσουμε όλους αυτούς ε, τους συλλόγους. Ο Νίλ είναι υπεύθυνο, ίσως μπορεί να σας πει δύο λόγια γι' αυτό, γιατί οργανώνουμε και ένα τουρνουά τον Ιούνιο και θα καλέσουμε όλες ε, τις ομάδες, ε, όλοι ε, στους συλλόγους που έχουν τις πρωτοβουλίες και θα κάνουμε μικτές ε, ομάδες, θα έχουμε πέντε πρόσφυγες και πέντε ε, παίκτες του συλλόγου και θα διασφαλίσουμε ότι μπορούν να παίξουν όλοι μαζί όπως κάνουμε και εμείς στο δικό μας σύλλογο. Πέρσι ήμασταν τυχεροί γιατί μας επισκέφθηκαν δύο επίτροποι, ο κύριος Αβραμόπουλος που είναι υπεύθυνο για τη μετανάστευση και ο επίτροπος αρμόδιος για τον αθλητισμό ο κύριος Τίμπορ Ναύρατσισκ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια υποστήριξη. Βλέπετε ότι έχουμε και κάποιους χορηγούς, όπως είναι το Ίδρυμα της ΟΕΦΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Ρουαμπουντάν, όπως είδατε. Έχουμε λοιπόν διάφορους πρωταγωνιστές ε, και από την κοινωνία των πολιτών, δημόσιες αρχές, ιδιωτικούς φορείς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό γιατί διαφορετικά δεν μπορεί κάποιος από μόνος του να φτιάξει ένα αξιοπρεπές project. Και ερχόμαστε στην τελευταία διαφάνεια. Τι ακολουθεί. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το δικό μας ε, μικρό project αποτελεί μέρος της διαδικασίας ένταξης των προσφύγων. Ο συνάδελφος θα μιλήσει γι' αυτό σε ένα λεπτό, αλλά είναι σημαντικό όλοι οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν να συμμετέχουν και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα, δημόσιες αρχές, να συνεργαστούν και να υπάρχει και ένα όραμα για να προσπαθούμε να βρούμε λύση για τους πρόσφυγες αυτούς. Γιατί όταν ε, συζητούμε μαζί τους, μας λένε ότι θέλουν να μείνουν εδώ, έχουν μακρύ δρόμο να διανύσουν, χρειάζεται πολύ υπομονή και χρειάζεται και δημόσια κονδύλια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διαφορετικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε κάποιες προϋποθέσεις ε, για να πετύχει το project, το περιβάλλον του καταρχήν. Ε, έχουμε έναν ομιλό που είναι πολυπολιτισμικός. Αυτό μας βοηθάει να έχουμε ένα τέτοιο project, διαφορετικά δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το πετύχουμε. Σε κάποιες άλλες τοποθεσίε μπορεί να είναι πιο δύσκολο να έχει ένα τέτοιο project. Και τα αριθμητικά στοιχεία, οι αριθμοί είναι σημαντικοί. Δεχόμαστε 6 με 10 πρόσφυγε την ημέρα. Δεν μπορεί να έχει πάρα πολλού. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Γκρέγκορη. Λοιπόν, ονομάζομαι Γκρέγκορη Μπλουικ, είμαι και ε, διευθυντής ενός ε, κέντρου ανηλίκων στο Σαν Πιά στις Βρυξέλλες ε, το κέντρο στο οποίο φτάνουν οι νέοι και τους οποίους φιλοξενούμε είναι η πρώτη επίσημη τους διεύθυνση. Μένουν σε εμά τέσσερις εβδομάδες, όσο χρειάζεται δηλαδή για να καταγράψουμε ένα προφίλ του νέου, έτσι ώστε σε μια δεύτερη φάση να προχωρήσει σε κάποιες δομές που συνάδουν με το προφίλ στο οποίο έχουμε καταλήξει. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος, χωρίς να μιλήσω πολύ γρήγορα. Ε, οι νέοι που ζουν στο Βέλγιο είναι, είναι περίπου 500 νέοι έρχονται κατά, κάθε μήνα, 520. Είναι ασυνόδευτοι ανήλικες, οι εθνικότητες που εκπροσωπούνται είναι το Αφγανιστάν, η Ερυθρέα πιο συχνά και η, Γουινέα. Ε, οι νέοι αυτοί Εξαρτάται βέβαια και από τη χώρα που προέρχονται, αλλά ας πούμε για τους Σύριους ε, έχουμε 90%, για τους Αφγανούς 70% είναι νέοι που έχουν την δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να παραμείνουν ε, στο βελγικό έδαφος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε. Ε, η ιδιαιτερότητα της υποδοχής μας εξαρτάται από την σταθερότητα και την ασφάλεια που προσφέρουμε στους νέους μας. Ε, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αισθάνονται ασφαλείς ε, τα, τα παιδιά που έρχονται, ασφαλεί τα παιδιά που έρχονται, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν καλές προθέσεις που κινούνται γύρω από την, από τα παιδιά αυτά. Έχουμε στο κέντρο αυτό έχουμε μια, ένα μηχανισμό συνοδείας αν θέλετε σε τρεις ε, φάσεις. Ε, ε, η πρώτη φάση αφορά το σεβασμό του νόμου, το σχολείο, η θρησκεία και δημιουργούμε έναν καμβά αν θέλετε, ένα πλαίσιο που δεν, το οποίο δεν μπορούμε να παρακάμψουμε και γίνεται και με κάποια προβολή και στο μέλλον χάρη στις ευρωπαϊκούς πόρους ε, έχουμε ένα, ένα πρόγραμμα ανταλλαγών. Ε, αυτό το οποίο θέλω στο κέντρο μας είναι να επωφελούνται όλοι οι νέοι. Ε, θέλω οι, οι ας πούμε, να μάθουν στους Αφρικανούς να παίζουν κρίκετ ε, χαίρομαι όταν οι Αφγανοί, οι Τσετσένοι, οι Σύριοι μαθαίνουν ποδόσφαιρο από τους Αφρικανούς. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσφέρουμε ε, δραστηριότητες ε, στους νέους που φιλοξενούμε, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα πεδίο ελευθερίας και ανταλλαγών, να, να ε, ζήσουν πράγματα τα οποία δεν προέρχονται από τη δική τους κοινότητα, όχι μονάχα στον αθλητισμό αλλά και στο φαγητό. Δηλαδή θέλουν, θέλουμε τα οι νέοι να δοκιμάζουν φαγητά τα οποία προέρχονται από άλλες χώρες και όχι από τις δικές τους. Ε, οι, νέοι που φιλοξενούμε έχουν καταλήψει τη χώρα τους. Αυτό είναι ένα γεγονός. Έχουν φτάσει σε εμά. Είναι επίσης ένα άλλο γεγονός. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η αρχή μιας διαδικασίας εδώ στο Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να συνοδεύουμε τους ε, νέους ε, και θα πρέπει να τους στηρίζουμε σε αυτά τα πρώτα βήματα τα οποία γίνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. όλες και όλους εσάς για αυτό το έργο που επιτελείται και το οποίο είναι έμπνευση για όλους. Η ενσωμάτωση δεν είναι και κανένα μικρό πράγμα και η νομοθεσία για το άσυλο είναι πολύ σημαντική, που τη συζητούμε άλλωστε όλη την ημέρα, αλλά και το να κατανοήσει κανείς ποιες είναι οι προκλήσεις της υποδοχής ανθρώπινων όντων στην κοινωνία μας, στις κοινωνίες μας, στις οικογένειες και ούτω καθεξής. Εγώ πιστεύω ότι οι εθνικοί βουλευτές θα πρέπει να προσέλθουν να συζητήσουμε σε μια συνάντηση και για την ενσωμάτωση με ανταλλαγή εμπειριών είναι νομίζω κρίσιμο να συμβάλλουν με την εμπειρία τους και οι εθνικοί βουλευτές. Τι σημαίνει δηλαδή επιτόπου η προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσίαση της προσπάθειάς σας. Έχετε και τα σχετικά φυλάδια τα οποία μπορείτε να ε, προμηθευτείτε έξω από την αίθουσα. Όντως είναι παράδειγμα που εμπνέει και άλλους ανθρώπους και οι πρόσφυγες συμβάλλουν στην ζωή των κοινωνιών. Νομίζω ότι έχω δίκιο που το λέω αυτό. Και ορισμένα από τα νεαρά παιδιά που έρχονται σήμερα εδώ στην Ευρώπη μπορεί αύριο να είναι οι αστέρες του ε, ποδοσφαίρου ή των άλλων αθλημάτων. Έχω την αίσθηση, λέει ο πρόεδρος, ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ. Νι, θέλετε να πείτε τίποτα. Θέλετε να ακούσετε κι άλλα. Αν η Κορνέλη ενδιαφέρεται να ακούσει κι άλλα, τότε μου αρκεί αυτό. Ορίστε, αρχίστε. Νόμιζα ότι μπορούσαμε να τελειώσουμε, αλλά ναι. Μπορεί να μιλήσει και κάποιο που να μην είναι λευκό. Μην πάρετε στραβά τα λεγόμενά μου, αλλά. Αυτό που λείπει εδώ είναι και ο πρόσφυγας, ε. Δεν θέλω βέβαια να επικρίνω κανένα, αλλά θα ήταν καλό αν είχαμε και τη φωνή ενό πρόσφυγα. Δεν είμαι πρόσφυγας. Ο πρόεδρος, ε, ήθελα να το πω αυτό. Δεν είμαι πρόσφυγας, είμαι μετανάστης. Ε, αλλά μέχρι εκεί φτάνουμε. Γεια σας. να έρθω λίγο σε αυτά που είπε ο Μπέντζαμιν. Βλέπω τον Μπέντζαμιν πώς δουλεύει με τα διάφορα παιδιά στο, στην ομάδα, στην ποδοσφαιρική μας ομάδα. Όταν έρχονται τα παιδιά στην ομάδα, έρχονται σε ομάδες γιατί πρόκειται από διαφορετικές χώρες, μιλούν διαφορετικές γλώσσες και έχουν και διαφορετικά χρώματα επιδερμίδας, να το πω έτσι, μιας και αυτά λέγαμε πριν με τον πρόεδρο. Ένα πράγμα που ξεπηδά είναι ότι όταν είναι στο γήπεδο, αν φύγουν από τη μέση όλα αυτά τα εμπόδια και πάνε οι άνθρωποι αυτοί να παίξουν ποδόσφαιρο, κρίκετ, βλέπουμε ότι τα παιδιά τα ξεχνούν όλα. Όλες τις διαφορές που τα χωρίζουν στη, στη ζωή τους. Και θέλω να δούμε μια κατάσταση. Αρχίσαμε νομίζω πριν από δύο εβδομάδες, Τετάρτη, είχαμε ομάδες από τη μια τους Αφγανούς και τους μαύρους Αφρικανούς από την άλλη και στο γήπεδο ένας Αφγανός ε, υπέστη ε, φάουλ, έπεσε. Ένας από τη μαύρη ομάδα ήρθε να τον βοηθήσει, να σηκωθεί. Ήρθε το μαύρο παιδί να βοηθήσει τον Αφγανό. Ε, μετά από την συνάντηση. Εγώ βρίσκω ότι είναι μαγική αυτή η σχέση που αναπτύσσεται. Έστω και για μια στιγμή υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος, ο δεσμός. Είναι μια στιγμή η οποία αλλάζει όλη την κατάσταση στον κόσμο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο αρκετά, αρκετά, αρκετή συζήτηση προκαλέσαμε. Τώρα νομίζω εξήγησα αυτά που ήθελα. κατάλαβα, καταλάβατε τι θέλω να πω. Μην φοβάστε. Την αλήθεια λέω. Όταν μιλείτε για empowerment, για ενδυνάμωση, ε, πρέπει να είναι και οι άνθρωποι αυτοί που λογαριάζεις να ενδυναμώσεις παρόντες. Ναι, είχαμε, είχαμε και τον σκοπό να φέρουμε και μερικούς από τους πρόσφυγες να τους φέρουμε εδώ. Να δείτε δηλαδή και ε, μαζί τους και γιατί μιλούμε, αλλά είναι δύσκολο. Διότι δεν μένουν πολλοί στα κέντρα, θα πρέπει να μιλούν γαλλικά ή αγγλικά για να καταλαβαίνουν και να τους καταλαβαίνετε. Και μάλλον δεν θέλατε να είναι και βαρετή η συνεδρία, έτσι δεν είναι. Καλά, με την επόμενη φορά φέρουμε μερικούς. Θέλετε εσείς να πείτε κάτι και μετά ολοκληρώνουμε. Καλησπέρα Σα. Ήθελα απλώ να πω την δική μου εμπειρία μέσα στα πλαίσια αυτού του project. Προσπαθούμε να τους ε, μάθουμε κάποιες βασικές έννοιες των γαλλικών. Προσπαθούμε να τους εξοικειώσουμε με την ε, το πώς λειτουργούν ε, οι Βρυξέλλες, ε, το Βέλγιο, τι είναι θεσμοί λίγο πολύ δηλαδή, γιατί είναι και χώρα που τους ε, φιλοξενεί και συζητώντας μεταξύ, μαζί τους προσπαθούμε να βρούμε κάποιες γέφυρες που να μας ενώνουν. Συζητάμε για το φαγητό, για το κλίμα, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έχουν δει ποτέ τους χιόνι, ας πούμε, και τους ενθουσιάζει ή τους ε, εξάπτει την φαντασία και την περιέργειά τους. Ε, συζητάμε και κάποια θέματα που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπήκανε στο τραμ, ας πούμε, που δεν είχαν ποτέ ποτέ τους. Ε, και βέβαια ένα σίγουρο θέμα συζήτησης είναι ο αθλητισμός. Τώρα, στους, υπάρχουν και κάποιοι περιερισμοί. Το ένα είναι ότι αλλάζει ο αριθμός, αλλά και οι νέοι αυτοί καθεαυτοί από εβδομάδα σε εβδομάδα προσπαθούμε να τους ε, γνωρίσουμε μεταξύ τους, αυτούς που έρχονται από την Αφρική, αυτούς που έρχονται από το Αφγανιστάν κτλ. Βέβαια το πρόβλημα είναι η γλώσσα επικοινωνίας. Κάποιοι γνωρίζουν κάποια γαλλικά ή αγγλικά ή γερμανικά, κάποιοι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα, καμία ευρωπαϊκή γλώσσα και προσπαθούμε από την ομάδα ε, που έχουμε ας πούμε, να έχουμε κάποιον Αφγανό ο οποίος μιλάει παστούν να λειτουργεί σαν διερμηνέας ε, με αυτό τους που δεν μιλάνε καμία ευρωπαϊκή γλώσσα. Πάντως για μένα αυτή η εμπειρία οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θεωρώ ότι ε, εμπλουτίζει την προσωπικότητα της τη προσωπικότητα όλων μα. Και τέλο πάντων ε, ήταν και πάρα πολύ ωραίοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνε που παρακολούθησα. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώ ε, η οικοδόμηση εμπιστοσύνη και το θέμα τη γλώσσα είναι στοιχεία πολύ σημαντικά για την ένταξη. Σα ευχαριστώ όλου για αυτό το εμπνευστικό project και είναι τόσο εμπνευστικό που σας επισκέφθηκαν και δύο επίτροποι. Είναι προφανώς ένα πολύ καλό το project αυτό για τους νέους πρόσφυγες. Σας ευχαριστούμε και που δεχτήκατε να έρθετε εδώ σήμερα και να μας δώσετε αυτά τα θετικά μηνύματα. Κάποιοι μας παρακολουθούν και μέσω του διαδικτύου. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ε, για το έργο σας, σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ και μας δώσετε αυτό το πολύ θετικό παράδειγμα. Και φυσικά που μπορούμε θα σας βοηθήσουμε στο μέλλον, συνάδελφοι. Ιδίω ε, όσοι μείνατε μέχρι το τέλος, σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας συνεισφορά στη διάσκεψη και ευχαριστώ όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και το προσωπικό για τη δουλειά του σήμερα. Θα δημοσιεύσουμε και τα αποτελέσματα των workshop και των ε, υπολείπων ε, συζητήσεων. Σας ευχαριστώ όλους ε, για την παρουσία σας και τη συνεισφορά σας.